Je de ε, Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, θα έλεγα το απόγευμα που μας περιμένει. Θα ακούσουμε και τον κύριο Μπάλκο από το ελεγκτικό συνέδριο. Θα υπάρξει επίσης μια ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Γενικό Διευθυντή κ. Λεμέτρ της Βέγγια. Να σας ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια των συντονιστών, της συνεδρίασης των συντονιστών, αποφασίσαμε να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα πάνω στην ε, μεγάλη καταστροφή στις αντίλες ε, με τον τυφώνα Ήρμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μια ανακοίνωση γύρω από το θέμα αυτό στο Στρασβούργο και το αίτημά μας σύνεπως θα ικανοποιηθεί. Λεπτομέρειες τώρα για την οργάνωση της ημερήσιας διάταξης θα σας δοθούν μέσω mail. Κύριε Λάντισλαβ Μπάλκο, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Η παρουσία σας εδώ στην Επιτροπή Ρέγγι είναι για μας ε, ιδιαίτερα σημαντική. Τακτικά το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ε, χορηγεί τις εκθέσεις που είναι η βάση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να χορηγήσουμε την απαλλαγή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκτιμούμε ιδιαίτερως και τις ε, ειδικέ εκθέσεις που εκπονείται εδώ και αρκετά χρόνια και που περιλαμβάνουν πολύ σημαντικά στοιχεία για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, γιατί έτσι μπορούμε και αξιολογούμε την εφαρμογή ε, των πολιτικών συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης στο σύνολο των κρατών μελών. Και επίσης, τα στοιχεία της έκθεσής σας είναι πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας. Ευελπιστώ λοιπόν ότι και μετά την ε, σημερινή ακρόαση η σχέση μεταξύ τη, της ε, δικής μας Επιτροπής και του Ελεκτικού Συνεδρίου θα συσφιχθούν έχετε εκπονήσει και ειδική έκθεση για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και μάλιστα μερικοί από εμά είμαστε στις ε, σχετικές διαπραγματεύσεις του κανονισμού. Γι' αυτό και περιμένουμε με ανυπομονησία την παρουσίαση της ειδικής σας έκθεσης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ε, ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου με αριθμό 2 του 2017 για τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2020 των συμφωνιών εταιρική ε, ε, σχέσης και των προγραμμάτων συνοχής. Μερικοί ήταν παρόντες και στην παρουσίαση που έκανα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 26 Ιουνίου και εκτιμώ ιδιαίτερως την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε, είχαμε τον κύριο Πυρίνσκι, τον αρμόδιο συγκεκριτή της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού και ευχαριστούμε για τα εύστοχα και τα αξιόλογα σχόλιά του τον ε, κύριο Βόν. Η σημερινή μου παρουσίαση αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Ελεκτικού Συνεδρίου για στενή συνεργασία με τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικά για θέματα που ενδιαφέρουν και τους δύο. Γι' αυτό και κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε την παρουσίαση όχι μόνο στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, αλλά και στις επιμέρους κοινοβουλευτικές επιτροπές. Στην ειδική μας έκθεση 2 του 2017 εξετάσαμε το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλέ διαπραγματεύσει των συμφωνιών εταιρική σχέση για το 2014-2020 και των επιχειρησιακών προγραμμάτων προκειμένου ε, να έχει πιο αποτελεσματική στόχευση των κονδυλίων της συνοχής και δαπάνη τους με τρόπο που θα εξυπηρετούν τη στρατηγική του 2020. Ε, και εξετάζουμε το κατά πόσο δικαιολογούνται οι παρεμβάσεις ό,τι αφορά τα αποτελέσματα και τις επενδυτικές ανάγκες και κάποια αξιολόγηση των αποδόσεων και το κατά πόσο συνέτρεχαν όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Και μάλιστα θα ακολουθήσει και δεύτερη έκθεση για τις ε, εκ των προτέρων και για το ε, αποθεματικό της απόδοση των επιδόσεων θεωρούμε ότι είναι καινοτόμο μέσο, αλλά όχι αρκετά αποτελεσματικό μέχρι στιγμής. Η δεύτερη έκθεση θα υποβληθεί στην τακτική διαδικασία που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός ο κανονισμός, ο αρμόδιος δημοσιονομικός κανονισμός, τη διαδικασία με τις κατέρωθαν ακροάσεις, κατά αντιπαράθεση, και επίσης μετά τη δημοσίευση ε, είμαι πρόθυμος να έρθω και να σας την παρουσιάσω και τη δεύτερη έκθεση, να το κρίνετε σκόπιμο. Τώρα να επισέλθω σε λεπτομέρειες για την ουσία της πρώτης μας αυτής έκθεσης, της του 2, 2017. Η Συμφωνία Εταιρική Σχέση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των κρατών μελών είναι στρατηγικά επενδυτικά σχέδια στα οποία τα κράτη-μέλη ε, επισημαίνουν τι εθνικέ του ε, προτεραιότητε δαπανών για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία σε μία επταετή περίοδο. Και μάλιστα οι διαπραγματεύσει έγιναν το 2014 και μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύτηκε 387 επιχειρησιακά προγράμματα για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Κοινωνικό Ταμείο με βάση αυτές ε, τις διαπραγματεύσεις και τα επιχειρησιακά προγράμματα. Επίσης, ε, στην, στον ε, έλεγχό μας κάνουμε και μια ανάλυση του χρονοδιαγράμματος, στον οποίο έγιναν οι διαπραγματεύσεις με βάση τις ιστορικές διαδικασίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναλύσαμε ε, εμβριθώς τις, εταιρικές, ε, τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 14 ε, επιχειρησιακά προγράμματα για ε, πέντε κράτη-μέλη, Ισπανία, Ιρλανδία, Κροατία, Πολωνία και Ρουμανία, καθώς και πραγματοποίησαμε και μια επίσκεψη Δανία, συνεντεύξεις με προσωπικό και υπαλλήλους των κρατών μελών και των μόνιμων αντιπροσωπιών και είχαμε και διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής και περιφερειακής συνοχής. Γενικώ βρήκαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αποτελεσματικό τρόπο διαπραγματεύτηκε τη Συμφωνία εταιρική σχέση και τα επιχειρησιακά προγράμματα 2014-2020 σε ό,τι αφορά τη συνοχή. Ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη εντός των κανονιστικών προθεσμιών. Ε, επικέντρωσε την χρηματοδότηση στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και ε, εξασφάλισε μια πιο στιβαρή ε, λογική παρέμβαση στα επιχειρησιακά προγράμματα. Δεν κατάφερε όμως ε, να εναρμονίσει την δημοσιονομική παρακολούθηση μεταξύ των κονδυλίων και της εξασφάλισης μιας σωστής καθορισμού των δικτών επιδόσεων για τις εκροές και τα αποτελέσματα. Αυτό, αυτό είναι μια σημαντική συνάθρηση και σύγκριση των δικτών ε, και των στοιχείων επιδόσεων μεταξύ των προγραμμάτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, επιπλέον στοιχεία, γιατί ο υπερβολικά μεγάλο αριθμό δικτών επιδόσεων και τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται ε, δημιουργούν διοικητικό άγχο. Τώρα, το κανονιστικό νομοθετικό πακέτο τη Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Συνοχή 2014-2020 υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2013, δηλαδή ένα πεντάμινο αργότερα από ότι στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Παρ' όλα αυτά τα κράτη-μέλη επέβαλαν όλες οι συμφωνίε εταιρική σχέσης εμπρόθεσμα και κατά μέσο όρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τι ενέκρινε μέσα σε πέντε μήνες, ε, ένα μήνα νωρίτερα από ότι τα εθνικά πλαίσια ε, στρατηγικής αναφοράς σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ήδη το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ανεπίσημες διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη και ε, ε κάτι καινούριο εξέδωσε ε, και έγραφα θέσεων με ανάλυση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη καθώς και πρόοδο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των στόχων του 2020 και τις ε, σημαντικότερες προτεραιότητες για χρηματοδότηση. Τα περισσότερα άλλα στα σχέδια επιχειρησιακών προγραμμάτων υπευλήθησαν από τα κράτη-μέλη έγκαιρα και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός των προθεσμιών και σε συγκρίσιμο χρονικό διάστημα σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Και μάλιστα διαπραγματεύσει των επιχειρησιακών προγραμμάτων μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κρατών μελών ήταν πιο δύσκολε και απαιτητικέ από τι προηγούμενε περιόδου. Και αυτό γιατί κάποια συμπληρωματικά κριτήρια όπω των προτέρων ερεσιμότητε ή η απέτηση να υιοθετηθεί μια πιο ε, ρητή λογική παρέμβαση. Κάποια προβλήματα επίση ε, τεχνολογίας των πληροφοριών απέτησαν περισσότερου γύρου εγκρίσεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αρχικά ε, σχέδια. Με βάση τις πρώτες αυτές ε, παρατηρήσεις συστήνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει τις νομοθετικές προτέσεις για την περίοδο μετά το 2020 εγκαίρως, ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος για τις νομοθετικές αρχές να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις. Δεύτερον. Όσον αφορά την εστίαση των δαπανών στους προτεραιότητες της στρατηγικής 2020, βλέπουμε πως η Συμφωνία Εσωτερικής Σχέσης είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για να διαφυλάξουμε την χρηματοδότηση για τους θεματικούς στόχους και τις προτεραιότητες που στηρίζουν τις, ε, τους στόχους της στρατηγικής και βεβαίως όλα αυτά καλύπτουν όλες τις ουσιαστικές πτυχές και παρέχουν μια διάγνωση των αναπτυξιακών αναγκών και των προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις. Οι απαιτήσει αυτές ε, κατά κανόν ε, ήταν κάτι το οποίο καταφέραμε και να ξεπεράσουμε. Δεδομένης δε, δεδομένου του γεγονότος ότι η επίτευξη των στρατηγικών αποτελεσμάτων σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σημαντική συνεισφορά από του εθνικού προπολογισμού. Προσπαθήσαμε να υπάρξει μια βελτίωση της γενικότερης δυνατότητας οικονομικής διαχείρισης από τα κράτη-μέλη. Επίσης, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη ανέπτυξαν επιτυχώς μια πιο εύρωστη λογική παρέμβαση. Αλλά βέβαια οι πληροφορίε τα επιχειρησιακά προγράμματα καμιά φορά δεν ε, συνάδει με αυτήν που υπάρχει στις ε, συμφωνίες εταιρική ε, σχέσης και για τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία χρησιμοποιούν παρεκκλήσεις συχνά δεν επιτρέπεται να υποληθεύσουμε εάν υπάρξει αυτή η θεματική συγκέντρωση. Με βάση αυτά εμείς προτείνουμε τα κρατη να δίνουν στην Κομισιόν τις πληροφορίες που χρειάζεται για να μπορεί να παρακολουθεί την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις θεματικής ε, συγκέντρωσης. Ε, επίσης θα πρέπει η Κομισιόν ε, να εξασφαλίζει ότι θα γίνεται σεβαστή η δεσμευσή των κονδυλίων. Και τώρα να έρθω στο σημαντικότερο θέμα της έκθεσής μας, την πολυπλοκότητα του προγράμματος 2014-2020 ε, που προκύπτει από διάφορους παράγοντες. Τον αριθμό των προτεραιοτήτων όπως το έχουν καθορίσει τα κρατημέλη, ο αριθμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν αλλά και ο αριθμός ε, των κατηγοριών περιφερειών που καλύπτονται από τα επιχειρησιακά προγράμματα εδώ πέρα. Θα πρέπει να δείτε ακριβώς ε, το τρισδιάστατο αυτό σχεδιάγραμμα που υπάρχει στην έκθεσή μας που υπάρχει ακριβώς στην, στο παρατήμα 3 στην σελίδα 89 της έκθεσής μας και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι αυτό δεν μπορούμε να το πούμε απλοποίηση. Επιπλέον, η προσέγγιση στην ε, χρηματοοικονομική παρακολούθηση των επενδύσεων διαφέρει μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης η σχέση μεταξύ των δράσεων και της χρηματοδότησης δεν είναι άμεση, ενώ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τα πεδία παρέμβασης ευθυγραμμίζονται πλήρω με τις προτεραιότητες επενδύσεων και κάθε προτεραιότητα είναι ένα πεδίο παρέμβασης, ενώ στο ΕΤΠΑ το ίδιο πεδίο παρέμβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές επενδυτικές προτεραιότητες. Έτσι, δεν μπορεί να παρακολουθηθεί σωστά η πρόοδος, καθώς δεν θα είναι σαφές πόσα κονδύλια πήγαν για την εφαρμογή των επενδυτικών προτεραιοτήτων που θα στηρίξει το ΕΤΠΑ. Συνολικά, όταν μιλάμε για τις διαφορές μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, θα πρέπει να δείτε το την εικόνα 15 στην σελίδα 74 που είναι ενδεικτική. Βλέπετε ότι για το ΕΚΤ υπάρχουν πολύ περισσότερα ισχυρά σημεία από ό,τι αδυναμίες και αντιστρόφως. Οπότε, κοινοί δείκτες ε, αποτελεσμάτων υπάρχουν μόνο για το ΕΚΤ και τα κράτη-μέλη έχουν συγκεκριμένους δείκτες αναπρόγραμμα, σχεδόν 3.000 τέτοιους δείκτες ε, για το ΕΤΠΑ και σχεδόν 2.000 για το ΕΚΤ. Αυτό αυξάνει κατά πολύ τον αριθμό των δικτών που πρέπει να προκληθούνται και έτσι δεν θα έχει κάποιο νόημα η σύγκριση και η συλλογή των δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψη δε το κόστος συλλογής αυτών των δεδομένων θεωρούμε ότι είναι πολύ υψηλός ο αριθμός των δικτών απόδοσης και δεν υπάρχει ένας κοινός ορισμός ε, του αποτελέσματος και της εκροής. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι περισσότερα και καλύτερα δεδομένα θα μπορέσουν να ανοίξουν τον δρόμο για έναν με βάση την απόδοση μετά το 2020. Με βάση λοιπόν αυτά προτείνουμε η Κομισιόν να καταλήξει σε κοινή ορολογία για τα αποτελέσματα και τις εκροές και να προτείνει να περιληφθεί στον δημοσιονομικό κανονισμό της Ένωσης για την περίοδο μετά το 2020. Προτείνουμε αυτό να γίνει στην πρώτη μας γνωμοδότηση για το 2017 για την αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού. Επίσης θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση των δικτών ανά πρόγραμμα και των κοινών δικτών για το 2014-2020 για τις εκλογέ εκείνες ε, και τα αποτελέσματα εκείνα τα οποία είναι καλύτερα για να δούμε τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων της Ένωσης. Τα κρατημέλη δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τέτοιους δείκτες στην περίπτωση που δεν χρειάζονται ή στην περίπτωση που αλλάξουν τα προγράμματα όπως γίνεται ήδη στην πραγματική περίοδο. Όσον αφορά τον αντίκτυπο των προγραμμάτων, αυτός φαίνεται στις αξιολογήσεις ε, και αυτό απαιτεί να είναι διαθέσιμα τα δεδομένα για τις ε, συγχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις και βέβαια τα κράτη-μέλη συστηματικά θα συλλέγουν και θα στέλνουν τέτοια δεδομένα στις Κομισιόν. Όμως, οι ε, δείκτες του ΕΤΠΑ δεν καταγράφουν τα άμεσα αποτελέσματα αυτών των έργων και δεν θα είναι διαθέσιμη εκτός εάν τα κρατημέλη αποφασίσουν να συλλέγουν επιπρόσθετα δεδομένα εθελοντικά. Προτείνουμε λοιπόν η Κομισιόν να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών όσον αφορά την αξιολόγηση και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στο να ενημερώσουν τα σχέδια αξιολόγησης που περιλαμβάνουν αυτές τις αξιολογήσεις βέλτιστων πρακτικών. Τέλος, θεωρούμε ότι διαφορετικές απαιτήσει στους κανονισμούς τους ε, για τα αποτελέσματα τα οποία μόλις ανέφερα είναι μια μεγάλη αδυναμία στο τρέχον σύστημα. Ως συνέπεια, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα παρακολούθησης της απόδοσης για το κάθε ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική μεθοδολογία και τον υπερβολικά μεγάλο ρυθμό δικτών. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο διοικητικό βάρος, αλλά βεβαίως ε, απομένει να δούμε και πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. Οπότε Προτείνουμε η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα από τις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής και αξιολόγησης για συγκριτική ανάλυση της απόδοσης και όπου αυτό απαιτείται να προτείνει την συγκριτική αξιολόγηση για να διδαχτούμε από την περίοδο 2014-2020 επίσης ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί η έννοια του προπολισμού με βάση την απόδοση που σημαίνει ότι η αύξηση στους θα πρέπει να συνδέεται με αύξηση στα αποτελέσματα ή ε, στις εκροές ε, χρησιμοποιώντας δεδομένα με βάση το πραγματικό μοναδιό κόστος όπως αυτό ήταν στην περίοδο 2014-2020. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας θα συνοψίσω τον τίτλο αυτής της έκθεσης Κομισιόν. Αποτελεσματικά διαπραγματεύτηκε τη Συμφωνία Τερικής Σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα 2014-2020 για να στοχεύσει καλύτερα στις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020, αλλά έχουμε όλο και πιο πολύπλοκες διευθετήσεις, ε, κάτι το οποίο είναι αιτία ανησυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την λεπτομερή ανακοίνωση. Έχουμε μισή ώρα τώρα για συζήτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που θέλουν το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κύριε Μπάλκο και σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Είναι σημαντική η έκθεση. Χαίρομαι που επιβεβαιώνεται πως ε, οι συμφωνίες σχέσεις ε, κρατών μελών και κομισιών κατέληξαν σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε κάποια προβλήματα βεβαίως ε, στο μέτωπο της ε, πληροφορικής ε, παραδείγματος χάρη. Έχουμε τις αρχές, τις διαχειριστικές στη Ρουμανία με τα γνωστά προβλήματα στον τομέα αυτών. Πώς θα μπορέσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι μετά το 2020. Θα κάνετε στοχευμένες συστάσεις στα κράτη-μέλη για να αποφύγουμε αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα μετά μιλήσατε πάρα πολύ σωστά για τα αποτελέσματα. Τι βεβαίω θέλουμε πράγματι να υπάρχει αξιολόγηση με βάση τα αποτελέσματα. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχω λοιπόν ένα ερώτημα. Σε ποιο βαθμό υπάρχει μια σχέση μεταξύ αυτών των δικτών και των στόχων ε, που καθορίζουν τις κοινέ διατάξεις. Και ποια είναι η σχέση επίσης ε, όσον αφορά τους δείκτες αυτούς και το αποθεματικό απόδοσης. Ελπίζω λοιπόν η Κομισιόν να αντιδράσει στην ε, έκθεσή σας με κοινού δείκτες για να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο συγκεντρωτικών στοιχείων και σύγκρισης για να μπορέσουμε πραγματικά να οδηγηθούμε στο σωστό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ, Κωνσταντς Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας ε, κύριε Μπάλκο για αυτή την πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Δεν έχω την έκθεση ε, μπροστά μου, οπότε όταν μιλούσατε για σελίδες ε, δεν μπόρεσα να δω αυτό το οποίο μας λέγατε, αλλά θα το κάνω. Κάτι άλλο. Τώρα έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τις συμφωνίες αυτές εταιρικής σχέσης το Κοινοβούλιο αποδώσει μεγάλη σημασία στο να ενισχυθεί η αρχή της ε, εταιρική ε, σχέσης. Είχαμε κάνει λοιπόν πάρα πολλές συζητήσεις ε, και ακούσαμε ότι η αρχή αυτή της εταιρική σχέσης δεν εφαρμόζεται τόσο απλά, αλλά σημαίνει λιγότερα δικαιώματα για τις τοπικές αρχές. Το ερώτημά μου είναι, εσείς ε, ψάξατε κάτι τέτοιο στην έκθεσή σας, έχετε σχετικές εμπειρίες, γιατί θεωρητικά η Κομισιόν θα έπρεπε να επιμείνει στην τήρηση της αρχής αυτής. Ήθελα λοιπόν να μάθω εάν έχετε κάτι σχετικά. Και μετά δικαίως είπατε ότι δεν σημαίνει πως οτιδήποτε έχετε γράψει είναι κάποια απλοποίηση, αλλά μπορείτε να, να μας μιλήσετε γενικά κάπως για την εξάντε αιρεσιμότητα, για το ότι βεβαίως οδήγησε σε χρονική καθυστέρηση όσον αφορά την υλοποίηση των πρώτων έργων. Εγώ θεωρώ παρόλα αυτά όμως πως αυτό ήταν σωστό γιατί θα αυξηθεί έτσι η ποιότητα των έργων, αλλά θα ήθελα να ακούσω την δική σας την εκτίμηση επ' αυτού. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε αν θα υπάρξει κάποια ενίσχυση της πολιτικής συνοχής ε, στο μέλλον και κάποια απλοποίηση της αιρεσιμότητας εξ άντε. Ευχαριστώ. Στο, εκ μέρους των Πρασίνων, ο κύριος Ροπέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και το ελεγκτικό συνέδριο. Πράγματι είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Έχει ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον και εγώ ως κάποιος ο οποίος θα ασχοληθεί ε, λίγο χρόνο με το να υποβάλω αιτήσει για έργα πλέον δεν μπορώ να αντιληφθώ τι γίνεται. Ας δούμε παραδείγματος χάρη το διάστημα αυτό το 2014-2020. Σήμερα είμαστε στον Σεπτέμβριο 2017. Τα έργα δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, οπότε δεν γίνονται πληρωμές. Όμως, η προθεσμία ήδη έχει περάσει στο δεύτερο μισό οι περιφέρειες δηλαδή επενδύουν ε, μόνο από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 80%. Αυτό σημαίνει ότι τα 2 τρίτα του χρόνου, 2-3 χρόνια δηλαδή 2-3 έτη, ναι, δεν μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις στα κράτη-μέλη. Τα κονδύλια λείπουν και απομένουν δύο χρόνια για να κινητοποιηθεί ολόκληρη η επένδυση. Αυτό σημαίνει ότι επιταχύνεται ο, ρυθμός, υπάρχει η απέτηση αυτή επιτάχυνσης και από εκεί προκύπτουν διάφορα λάθη και ελλείψεις. Οπότε σας ερωτώ, μήπως σκέφτεστε ότι ε, θα μπορούσαμε για την επόμενη περίοδο από το 2020 και μετά να ξεκινήσουμε τότε ε, με την εφαρμογή για να δούμε αμέσως τα έργα από το 2020 ή ε, θα προτείνετε κάτι διαφορετικό έτσι ώστε αφενός να έχουμε βιώσιμες επενδύσεις και αφετέρου να μπορέσουμε να κατευθύνουμε και επενδύσεις στην βιομηχανία, στη βιοτεχνία, όπου λείπουν οι επενδύσεις και αναζητούν αλλού τελικά επενδυτές ή επιχειρήσεις. Κατόπιν για τα προγράμματα και τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Συγκεκριμένα, σήμερα νωρίς το πρωί συζητήσαμε για τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν χώρες που δεν έχουν περιφέρειες. Ε, δηλαδή η Λιθουανία είναι μία περιφέρεια. Αλλά σε αυτήν την περιφέρεια υπάρχουν διαφορές. Αλλά δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για τις διαφορετικές περιοχές ε, μιας χώρας ε, για να λαμβάνουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Οπότε έχουν περισσότερες επενδύσεις οι πιο ανεπτυγμένες ε, περιοχές και βεβαίως οι άλλες μένουν πίσω. Ο κύριος Μάτο και μετά ο κύριος Πίρσεν που θα είναι και τελευταίος. κυρία Ευχαριστώ τον δόκτωρα Μπάρκο για την παρουσία του. Όπως μας είπατε ήδη, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κράτη-μέλη επιδιώκουν τις συμφωνίες ε, εταιρικής σχέσης όπως προβλέπονται από τις ε, αποφάσεις που είχαν ληφθεί στο παρελθόν. Υπάρχουν όμως κάποια κενά και κάποιοι σημαντικοί ορισμοί δεν έχουν γίνει αντικείμενο σωστού ε, συντονισμού και επικοινωνίας. Στις τελικές συστάσεις το ελεγκτικό συνέδριο λέγει αυτό που μας έχει πει επανειλημμένα ότι υπάρχει ανάγκη δηλαδή για μια νέα πρόταση για το 2020 από την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν έτσι ώστε να διαπραγματευθεί η Επιτροπή με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο <clears throat> το πλαίσιο αυτό και να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σε επίπεδο λειτουργικών προγραμμάτων και εταιρικών σχέσεων, συμφωνιών τα λειτουργικά προγράμματα της Νότιας Ιταλίας εγκρίνθηκαν ε, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2015, κάτι το οποίο επηρέασε και την ποσότητα και την ποιότητα της προβλεπόμενης δαπάνης. Στην ε, παρατήρηση 55 ε, κάνετε αναφορά σε πληροφορικά προβλήματα σε επίπεδο ηλεκτρονικής, πληροφορικής κτλ. για τον τομέα της κατάρτισης. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει η έκθεσή σας, χρησιμοποιείται ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς έχει πολλαπλές μορφές, 19 συγκεκριμένα, και γι' αυτό ακριβώς η επιθυμία μας για απλοποίηση των διαδικασιών δεν εξυπηρετείται. Πώς λύνεται το πρόβλημα αυτό και πώς σκοπεύεται σε επίπεδο λειτουργικών προγραμμάτων να προχωρήσετε. Το αίτημα αυτό αφορά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο το συνέδριο. Ευχαριστώ κύριε Σινίρσον. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά την προετοιμασία αυτή αυτής της περίοδου προγραμματισμού 2014-2020 εκπροσωπούσα μια περιοχή της Βορείου Σουηδίας που ήταν πολύ επικριτική για τον τρόπο που η Σουηδική κυβέρνηση διαπραγματευόταν τις συμφωνίες εταιρική σχέσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ερήμην των περιφερειών, χωρίς καμία εμπλοκή, καμία προσπάθεια ανάμειξης των περιφερειών. Ε, ερωτώ λοιπόν, εξετάσατε καθόλου αυτό ακριβώς το στοιχείο, κατά πόσο η, τα κράτη-μέλη εμπλέκουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ή έχετε προβεί σε κάποιες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι κάνατε συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά προς τα κράτη-μέλη έγιναν αντίστοιχε συστάσεις για περισσότερη εμπλοκή των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών. Για να προσθέσω κι εγώ λίγη δυσκολία στο έργο της απάντησε τόσο περίπλοκες ερωτήσεις. Ε, θα προσθέσω και τη δική μου ερώτηση και θα σας ενημερώσω ότι έχετε μόνο ένα δεκάλεπτο για να απαντήσετε. Στην έκθεσή σας επισημαίνετε ότι δεν υπάρχει κατά ανάγκη σύγκληση των επιδόσεων και των θεματικών στόχων. Ερωτώ λοιπόν, ποιοι είναι οι θεματικοί στόχοι που δεν έχουν υλοποιηθεί, που παρακάπτονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί μιλήσατε για το θεματικό στόχο της αηφόρου ανάπτυξης και τη μετάβαση σε μια οικονομία απαλλαγμένη από εκπομπές άνθρακα. 20% μάλιστα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, αφιερώνεται στην ε, επίτευξη αυτού του στόχου. Ε, παρακαλώ, έχετε ένα δεκάλεπτο για να απαντήσετε. Ελπίζω να καταφέρετε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις για να διαμορφώσουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Επιτροπής ε, για τις παρατηρήσεις τους. Έλαβα το λόγο 6-7 ευρωβουλευτές, κάτι που δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριος Μίλτεμπουργκ είπε ότι εσείς ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα επιστήσετε την προσοχή σε αυτά τα θέματα κατά την προετοιμασία του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά α, τις ερωτήσεις Ρόμπιν και άλλων, ίσως λύση καλύτερα να δώσει οι απαντήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η πλέον αρμόδια και όχι εμείς ως ελεκτικό συνέδριο εμείς ε, με βάση τα πορίσματά μας ε, ε, συντάξαμε έξι συμπεράσματα ενίδησης στάσεων και επαναλαμβάνω θα εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία με ακρόαση όλων των ενδιαφερομένων κατά την παράθεση και από το δικό μου επιτελείο Μπρανίσλαφ συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία όπου γίνεται αυτή η παρουσίαση κατά αφισβήτηση και υποβάλλονται ερωτήσεις στις οποίες δίνονται απαντήσεις. Ε, ο Μπέραντ Βίτκοπ επίσης ε, είναι σε θέση να σας ε, δώσει πιο σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες γιατί συμμετείχε σε αυτή την κατά την παράθεση διαδικασία. Ο Μπράνισλαφ. Ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω καταρχήν να απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά που υπευλήθησαν και δεν ξέρω αν ο Μπερνάρ θέλει να συμπληρώσει κάποιο στοιχείο. Καταρχήν, κύριε Φαν Μίλτεμπεργκ, μιλήσετε για τα θέματα τεχνολογίας των πληροφοριών. Ε, το ίδιο θέμα επισήμανε και ο Ευρωβουλευτής που έθεσε την τέταρτη ερώτηση. Δεν έχουμε ειδικέ στάσει ή συγκεκριμένε στάσει για τα προβλήματα τεχνολογιών τη πληροφορία που εντοπίσαμε. Αναφέρεται στην παράγραφο 55 της έκθεσής μας. Πάντως, ε, για την εξάντια ερεσιμότητα χρειάζονται συστήματα και ικανότητες στα κράτη-μέλη που περιλαμβάνουν και τα συστήματα πληροφορικής. Οπότε, ε, το επισημαίνουμε πάντως και στην επόμενη έκθεση που θα δημοσιευθεί στα τέλη του τρέχοντος ή στις αρχές του επόμενου έτους, θα αγγίψουμε περαιτέρω στο θέμα αυτό. Η δεύτερη ερώτηση του κ. Μιλτέμπερκ αφορούσε τους δείκτες που σχετίζονται με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Ε, είναι λοιπόν σαφής αυτός ο δεσμός, αλλά το πρόβλημα που εντοπίζουμε είναι ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των δικτών και μάλιστα είναι και περίπλοκοι οι δείκτες. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που καταμετρούν με διαφορετικό τρόπο το ίδιο πράγμα. Είναι πληθώρα των δικτών στα προγράμματα, κάτι που καθιστά δύσκολη τη συνάθρηση των στοιχείων και τη συγκριτική αξιολόγηση. Επισημάναμε λοιπόν αυτή την αδυναμία που οφείλεται στον υπερβολικά μεγάλο αριθμό των ε, ειδικών δικτών επιδόσεων. Η κυρία Κρέλ μίλησε για την αρχή της εταιρικής σχέσης και το κατά πόσο αποδυναμώθηκε από το γεγονός ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν αναμειχθήκαν δεόντως στις διαπραγματεύσεις. Το ίδιο η παρόμοια ζήτημα έθιξε και ο τελευταίος ομιλητής. Δεν επικρίνουμε αυτό το σημείο, δεν εγγύψαμε στην έκθεσή μας αυτό το θέμα του βαθμού ανάμειξης των τοπικών και περιφερειακών φορέων και αρχών, γιατί στη διαδικασία ανάθεσης σεβόμαστε την αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια να Επισημάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιο είναι αρμόδιος με βάση το εθνικό δίκαιο για το α ή το β πρόγραμμα ή το α ή το β κονδύλιο. Σε ό,τι αφορά την εξάντια, την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα, την εκ των προτέρων αιρεσιμότητε, αφορά δύο παραγράφους της έκθεσης και θα αναλυθεί πιο διεξοδικά στην δεύτερη έκθεση που από την επόμενη εβδομάδα θα, ξεκινήσει την, κατά την παράθεση διαδικασία, οπότε ίσως γίνουν κάποιες αλλαγές. Πάντως η βασική ιδέα είναι ότι η καινοτομία είναι κάτι θετικό, καλό, αλλά στην πράξη δεν βλέπουμε όλα τα αποτελέσματα, όλα τα θετικά της αποτελέσματα. Γιατί ελέγχθηκε το θέμα αυτό και αρχικά και το 2016, αλλά έκτοτε δεν έχουμε έλεγχο του κατά πόσο ισχύει ακόμη η εξάντε αιρεσιμότητα. Και ίσως αυτή είναι κάποια μορφή που ίσως αναλυθεί περαιτέρω στην δεύτερη, την επόμενη έκθεση που θα συντάξουμε σχετικά. Η τρίτη ερώτηση ήταν του κυρίου Ροπέ. Το αφορά τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Πάντα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος και τον έχουμε επισημάνει επανειλημμένος. Όσο πιο αργά ξεκινάει η διαδικασία, ε, τόσο χαμηλότερος είναι ο ρυθμός ε, απορρόφησης ή ε, εφαρμογής και υπάρχει και ο κίνδυνος διάπραξης φαλμάτων. Και αυτό το κίνδυνο το διατρέχουμε αυτή τη στιγμή λόγω της καθυστέρησης. Και αυτό λέμε και στην πρώτη μας σύσταση, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει εγκαίρω την νομοθετική βάση και επίσης να εγκρίνεται αυτή η νομοθετική πρόταση εγκαίρως και από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, το θέμα της εταιρική ε, σχέσης και των συμφωνιών εταιρική σχέσης είναι εθνική αρμοδιότητα. Το ε, κράτος μέλος με βάση το εθνικό δίκαιο θα επισημάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αρμόδια αρχή. Δεν μπορούμε εμείς ούτε δικαιούμαστε να υποβάλουμε επικρίσεις σχετικά στα κράτη-μέλη για χαμηλή εμπλοκή ε, των περιφερειακών αρχαίων. Ε συντομία παρακαλώ και μετά θα ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όντως ε, το συζητήσαμε το θέμα της ε, εταιρική σχέσης και τις ε, εταιρικέ σχέσεις που έχουν θεσπίσει τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη αυτών των συμφωνιών εταιρική σχέσης. Το έχουμε συζητήσει, αλλά δεν είναι και το κεντρικό θέμα του, ε, της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου, δηλαδή ανάλυση της αρχής της εταιρική σχέσης καθ' αυτής. Και παραλαμβάνω ότι δεν μπορούμε, είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε την ποιότητα της εταιρική σχέσης, γιατί μπορούμε να το αξιολογήσουμε ποσοτικά, αριθμό συνεδριάσεων, ανάμειξη εταίρων, αλλά η ποιοτική αξιολόγηση, η αξιολόγηση της ποιότητας της εταιρική σχέσης ε, ε, είναι ένα πιο απαιτητικό και δύσκολο ζήτημα γιατί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο δέσμευσης, την ανάληψη ευθύνης και αυτό είναι δύσκολο να καταμετρηθεί. Πάντως τα κράτη-μέλη που εξετάσαμε πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις για τις ε, εταιρικές σχέσεις και την ανάμειξη των αρμοδίων ενδιαφερομένων εταίρων. Ευχαριστώ. Je vous remercie. Je vous remercie pour ces éléments. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Οπότε παροτρύνετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συστήνετε στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία να υποβάλει την νομοθετική της πρόταση σε έφετο χρόνο, ε, εγκαίρος. Και συμφωνώ μαζί σας, όπως ε, συμφωνώ φυσικά και με την ε, ανάγκη της απλούστευσης. Απλούστευση, απλοποίηση και ταυτόχρονα έγκαιρη υποβολή της νομοθετικής πρότασης, ώστε να εγκριθεί και αυτή εμπρόθεσμα. Έτσι δημιουργούνται οι καλύτερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των μελλοντικών προγραμμάτων. Γνωρίζετε όμως τι δυσκολίες υπάρχουν και τι αβεβαιότητες ως προς το χρονοδιάγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζο, η κυρία Κατρίν, Κατρίν Ερστάλ, θα μας καθησυχάσει για το θέμα της στήριξης του χρονοδιαγράμματος. Παρακαλώ. Ναι, φυσικά και είμαστε παρόντες εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει το Ελεκτικό Συνέδριο για το ότι εντόπισε τους σωστούς στόχους και ε, διευκρίνησε ότι παρά την ε, περιπλοκότητα και τη δύσκολη κατάσταση λόγω της καθυστέρησης ε, του Πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, κατάφερε παρόλα αυτά να υιοθετήσει ε, τις συμφωνίε σχέσεις και τα επιχειρησιακά προγράμματα εγκαίρως και να καλύψει ε, τις καθυστερήσεις από νομική άποψη. Επίσης ε, χαίρομαι που και από άποψη διαδικασίας και από άποψη χρόνου ήμασταν εμπρόθεσμοι και γνωρίζετε τα πολύ σημαντικά στιβαρά προγράμματα που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τις προτεραιότητες της στρατηγικής του 2020. Θα ήθελα να σταθώ ε, σε κάποια ζητήματα. Βέβαια, πολλά από αυτά αφορούν το μέλλον και δεν είναι το αντικείμενο της ε, συγκεκριμένης έκθεσης και ναι και ο Γενικό Διευθυντή θα έρθει κάποια στιγμή στην Επιτροπή σα, μπορείτε να θέσετε εκεί ε, τι πιο στρατηγική φύσεω ερωτήσει σα. Εκεί θα συζητήσετε μαζί του και το θέμα του χρονοδιαγράμματος τη ε, της επόμενης πρόταση πρότασης για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Γενικό Διευθυντής μας είναι πλέον αρμόδιο να απαντήσει στις σχετικέ ερωτήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά του δείκτε δεν διαφωνούμε με το δικαστήριο ότι όντω ε, είναι πολύ άριθμοι οι δείκτες και μάλιστα αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τους ειδικού δείκτες των προγραμμάτων γιατί έχουμε εκατοντάδες προγράμματα και διαπιστώσαμε και εμείς ότι για παρόμοια θέματα έχουμε διαφορετικούς ειδικού δείκτες. Ε, επίσης εξετάζουμε με βάση αυτούς ε, το, το ύψος των κονδυλίων και ε, διερευνούμε κατά πόσο την επόμενη φορά θα μπορούσαμε να προτείνουμε πανευρωπαϊκούς α, δείκτες. Επίσης, αναφερθήκατε για δύο με τρία χρόνια σε ό,τι αφορά το επενδυτικό κενό. Ε, στην παρούσα δημοσιονομική περίοδο, με το σύντρία που θα προσθεθεί, θα έχουμε, έχουμε κοστά μας μία εξαιτία. Οπότε έχουμε αρκετό χρόνο. Αυτό βέβαια δεν μας κάνει να επαναπαυόμαστε. Αλλά αν εξετάσουμε τέσσερις συναπτές περιόδους προγραμματισμού, διαπιστώνουμε ότι είναι σταθερή η επενδυτική ροή. Γιατί ενώ μια επενδυτική περίοδος ξεκινά αρχικά με αργούς ρυθμούς, μια άλλη ολοκληρώνεται. Και το 2014, με βάση τις αρχικές μας προτάσεις, ε, τα περισσότερα 47% των κονδυλίων ε, ε, εκταμιεύτηκαν αργά στην περίοδο το 2012 και 2013, αλλά προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε σχετικά ομαλές επενδυτικές ώρες στις περιφέρειες. Επίσης, 40% είναι ε, ο συντελεστής ε, επιλογής, οπότε ε, είναι σημαντική δουλειά που γίνεται, απλώς δεν έχουν φτάσει ακόμη όλες οι πληρωμές. Τώρα, για τις περιφέρειες που δεν είναι περιφέρειες NATS 2, είναι και πάλι θέμα εθνικής απόφασης και εθνικής περιφερειακής πολιτικής. Εμείς ε, προβλέπουμε στήριξη, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τις δικές τους εθνικές περιφερειακές πολιτικές για να μπορέσουμε να τις στηρίξουμε. Και δεν μπορούμε να πιέζουμε τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν τέτοιες πολιτικές αν δεν τα επιθυμούν. Πάντως για τους δείκτες εν γέννη σας παραπέμπω στο άρθρο 16 ε, και στη σχετική έκθεση που υπευλήθη στην Επιτροπή και θετήθηκε τέλη του 2015 κατά το τέλος της περίοδου διαπραγμάτευσης για τα προγράμματα και βλέπετε ότι το ισχύον σύστημα δικτών είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, των προηγούμενων περίοδων ε, προγραμματισμού. Και έτσι ενημερώνονται οι φορολογούμενοι πολύ καλύτερα για το πώς δαπανώνται τα κονδύλια. Οπότε έχουμε καλύτερη καταμέτρηση της χρηματοδότησης και ε, εξακριβώνουμε κατά πόσο τηρήθηκαν οι υποσχέσεις. Και τώρα θα ξεκινήσουμε και εμείς την ενημέρωση για το πόσο οι δείκτες και οι στόχοι εφαρμόζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την παρουσία του και την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό που είπατε στην αρχή της συνεδρίασης. Φυσικά αρμόδια ε, είναι για το θέμα αυτό η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού που αναλαμβάνει τι ευθύνε τη, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τις υπόλοιπε, ε, τι ειδικέ κοινοβουλευτικέ επιτροπέ που ενδιαφέρονται για τις ε, ειδικέ σα εκθέσει. Και όλα αυτά θα συμβάλλουν ώστε να έχουμε καλύτερη χρήση και απόδοση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών κονδύλιων. Μια σύντομη διακοπή, δίλεπτη, περιμένοντας τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Λεμέτρ.

Bien. Nous poursuivons notre ordre du jour. Λοιπόν, επανερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ που θα πάρετε όλες τις θέσεις σας. Έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε σήμερα τον Γενικό Διευθυντή της DG Regio, τον κύριο Μάρκ Λεμέτρα. για την περιοδική ανταλλαγή απόψεων. Γνωρίζετε ότι ο Γενικός Διευθυντής είναι στη διάθεσή μας και μπορεί να απαντήσει και στο σύνολο των ερωτήσεων, αλλά θα πρέπει να οργανώσουμε κάπως τη συζήτηση και ε, με βάση τις ερωτήσεις οι οποίες είναι οι πλέον σημαντικές αν θέλετε και μετά και από κάποιες διευκρινήσεις τις οποίες μπορούμε να δώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνήσαμε ο, ε, Γενικός Διευθυντής να παρουσιάσει την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λεγόμενη ευφυή εξειδίκευση για την θέση σε εφαρμογή των ε, ενισχύ προγραμμάτων. Είμαστε πολύ κοντά δηλαδή ε, στην ακρόαση την οποία θέλουμε να οργανώσουμε με το συνέδριο, το ελεγκτικό συνόμι συνέδριο και με το θέμα για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τις καινοτόμες συγγνώμη, δράσεις σε αστικές περιοχές στα πλαίσια του ΦΕΝΤΕΡ. Όπως βλέπετε κύριε Λεμέτρο δεν θα αποφύγετε να δώσετε και πιο στρατηγικές απαντήσεις σε σχέση με το μέλλον της πολιτικής συνοχής, αν και γνωρίζουμε ότι κάποιες απαντήσεις δεν μπορούν να δοθούν παρά από την Επίτροπο Κρέτσου. Σας δίνω το λόγο λοιπόν και αμέσως μετά θα δώσω το λόγο στους συντονιστές και στα μέλη που έχουν ερωτήσεις να σας θέσουν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, αγαπητά μέλη. Θα ε, ήθελα να προσθέσω ένα πράγμα μόνο. στην ημερήσια ε, διάταξη που αναφέρατε και αυτό αφορά την επικοινωνία. Γιατί νομίζω πως είναι κατάλληλη στιγμή να κάνουμε έναν απολογισμό. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομος για να μείνει και χρόνος ε, για συζητήσεις πράγματι εγκρίναμε μία ανακοίνωση ε, για την έξυπνη εξειδίκευση, αυτή είναι η ουσία της έκθεσης, τον Ιούλιο. Νομίζω ότι κατά την άποψη της Επιτρόπου και της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, Περιφερειακής ε, Πολιτικής δεν είναι μια τυπική ανακοίνωση, είναι μια ουσιαστική, σημαντική και τολμώ να πω μια στρατηγική ανακοίνωση. Είναι νομίζω μια σαφής ένδειξη για το ότι η καινοτομία ήδη αυτή τη στιγμή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πολιτική αυτή και ο ρόλος της αυτός θα εδρεωθεί στο μέλλον. Και θα ξεκινήσω με τον απολογισμό αυτής της ανακοίνωσης. Και βεβαίως θα έλεγα πως ε, υπάρχει ακριβώς αυτό το μεγάλο επίτευμα της ε, πολιτικής ε, συνοχής ε, που είχαμε ακριβώς αυτή την επανάσταση των, πολιτι... των δημοσίων πολιτικών καινοτομία. Είχαμε ξεκινήσει το 2008-2009 κάπου εκεί σε ακαδημαϊκούς κύκλους και Δέκα χρόνια μετά η Ευρώπη ε, εφαρμόζει συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα και ε, μας παρακολουθεί ο υπόλοιπος πλανήτης. Ε, ενημερώθηκα σήμερα από έναν από τους πανεπιστημιακούς που επινόησαν την ιδέα σχετικά και όλα αυτά προέκυψαν χάρη στην πολιτική συνοχής και τον νέο μηχανισμό της εξάντε ερησιμότητας, ε, για να είμαστε ακριβείς. Γιατί ακριβώς αυτό ήταν από τους όρους για να διατεθούν τα κονδύλια της ε, συνοχής. Ε, έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα έλεγα, των δυνατοτήτων πίεσης που έχει αυτή η πολιτική και μόχλευσης. Επίσης είναι αξιοθαύμαστο ότι είναι μία από τις λίγες ε, αίρεσιμότητες ε, εξ άντε που γενικά αγκαλιάστηκαν θα έλεγα με μεγάλο ενθουσιασμό και χωρίς κανένα πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε πάνω από 120 τέτοιες ε, έξυπνες στρατηγικές Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν ε, έχουμε ακόμα ολοκληρώσει την επανάσταση αυτή. Βεβαίω, η άμεση ε, ανάγκη είναι το ότι μιλάμε για έγγραφα τα οποία εξελίσσονται και οι στρατηγικές αυτές χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες προκηρύξεις για έργα και αυτό είναι ευθύνη των διαχειριστικών αρχών σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί έχουμε πολύ σημαντικά ποσά βεβαίως, τα οποία πρέπει να διατεθούν στην καινοτομία ε, γύρω στα 70 δισεκατομμύρια στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο που ίσως ε, να το προσέξατε είναι σχεδόν ε, όσο το πρόγραμμα Horizon 2020. Και μετά βεβαίως υπάρχουν και κάποια στοιχεία στα οποία δεν ε, έχουμε, θα έλεγα, ακόμα φτάσει στις βέλτιστες συνθήκες όσον αφορά όλους τους δρόντες. Θα τρία στοιχεία βελτίωσης ε, στο προσεχές μέλλον που θα θέλαμε να δούμε. Το πρώτο είναι η ευρωστία των συστημάτων καινοτομίας στο περιφερειακό επίπεδο. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται πάντα στις ανάγκες και τις δυνατότητες των τοπικών οικονομιών. Είναι ζήτημα δομών, κινήτρων, προσέγγισης ε, στον ακαδημαϊκό κόσμο, στα πανεπιστήμια, σε επιχειρήσεις κτλ. Και βεβαίως ε, για να υπάρξει κάποια βελτίωση θεωρώ και πάλι ότι η πολιτική συνοχή έχει τα κατάλληλα εργαλεία. Οπωσδήποτε έχουμε τις ε, δυνατότητες μέσω της επανεξέτασης της ε, αιρεσιμότητας εξάντε να επιτύχουμε και κάποιες ουσιαστικές ε, διαρθρωτικές αλλαγές στα οικοσυστήματα αυτά θα έλεγα στην αρχή της επόμενης περίοδου. Αλλά ήδη από τώρα θα θέλαμε να υπάρξει κάποια θετική αλλαγή και για τον λόγο αυτόν έχουμε μια κοινή προσέγγιση με την Γενική Διεύθυνση Ερεύνης ε, και χρησιμοποιώντας μια δέσμη του ορίζοντα 2020 που αφορά ακριβώς την βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων καινοτομίας. Ελπίζουμε να σημειώσουμε ήδη σημαντική πρόοδο. Ο δεύτερος τομέας βελτίωσης, όπου η βελτίωση είναι ορατή, είναι η ανάγκη να υπάρξουν έξυπνες στρατηγικές καινοτομίες χωρίς εσωστρέφεια που θα υπάρχουν σε μία μόνο περιφέρεια δηλαδή και θα κοιτάνε προς τα μέσα αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικότητες της παγκόσμιας οικονομίας, ε, του πώς αναπτύσσεται μέσω μιας αλυσίδας προστιθέμενης αξίας και έξυπνες ε, στρατηγικές ε, εξειδικεύσεις που θα μας δίνουν την δυνατότητα να βρούμε κάποιους εταίρους για να συνεργαστούμε με τρόπο διαπεριφερειακό έχουμε δημιουργήσει. Κάποια αρχή έχουμε, παραδείγματος χάρη, τις ε, θεματικές πλατφόρμες. Αφορούν το βιομηχανικό μετασχηματισμό, την ενέργεια και τη γεωργία. Βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν ε, δίνει τις δυνατότητες στις περιφέρειες που θέλουν να κάνουν κάποιες κοινέ επενδύσεις, π.χ. για ένα έργο επίδειξης, για νέες ε, διαδικασίες παραγωγής, να συγκεντρώσουν τα λεφτά και να υλοποιήσουν αυτά τα έργα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη περίοδο, ειδικά, αλλά και στο άμεσο μέλλον, με την χρήση κάποιας ε, τεχνικής αρρωγής, αρωγής ε, που χρησιμοποιεί η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής ε, Ανάπτυξης για να κινητοποιηθούν έτσι αυτοί που πραγματικά θέλουν να συνεργαστούν. And I think Τέλος. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη εμπειρία πολιτικής για τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης ε, θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη αφετηρία για τις περιφέρειες εκείνες που βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο θα έλεγα όχι μεταβατικές περιφέρειες όπως λέμε αλλά α, περιφέρειες και οπωσδήποτε όλοι ξέρουμε τέτοιες, ε, οι οποίες λόγω διαφόρων αιτιών, π.χ. του ότι είχαν κάποιες ιστορικές βιομηχανίες, όπως παραδείγματος χάρη η χαλιβουργία, η φαντουργία, η παραδείγματο χάρη προσεχώς ε, η ξόριξη άνθρακα που κάποια στιγμή τις επόμενες δεκαετίες θα λήξει. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν μια μετάβαση, να αναπτύξουν νέους κλάδους της οικονομίας. Είναι μια τεράστια πρόκληση και παλεύουν περιοχές στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες βεβαίω για να κάνουν αυτή τη μετάβαση. Θεωρούμε ότι οι στρατηγικές και εξειδικεύσεις προσφέρουν μια καλύτερη αφετηρία από τα όσα είχαν μέχρι στιγμής επιχειρηθεί. Και εκεί πέρα ακριβώς ε, θέλουμε να υπάρξει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ίδιες τις περιφέρειες ε, που θα έχουν το ενδιαφέρον για να στηρίξουμε αυτό με όλα τα μέσα των ε, υπηρεσιών της ε, Κομισιόν ε, που θα μπορούσαν να έχουν εμπειρία και ακόμα και εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη εάν ε, αυτό απαιτείται. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά σημεία όπως τα βλέπουμε εμείς τα σημεία για τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά νομίζω ότι το βασικότερο μήνυμα εδώ πέρα είναι ότι είμαστε βαθύτατα πεπισμένοι ότι έχουμε εδώ πέρα κάτι το οποίο παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες για την Ευρώπη, για την πρόκληση του βιομηχανικού μετασχηματισμού, για το πώς θα διαχειθεί η τεχνολογική αλλαγή στους διάφορους κλάδους ε, στην Ευρώπη και άρα ε, αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε μακροπρόθεσμα και νομίζω πως έχουμε αυτήν την πεποίθηση γιατί βλέπουμε το πόσο ενθουσιοδός ε, έχει αγκαλιαστεί αυτό στο περιφερειακό επίπεδο και πώς έχει κινητοποιήσει τον κόσμο. Αυτά για αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα για την εφαρμογή του προγράμματος. Εκεί πέρα δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα θα έλεγα. Έχουμε λάβει τα τελευταία δεδομένα που μας έστειλαν τα κρατη τον μήνα Ιούλιο και δεν μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Όπως λέμε στα γαλλικά, έχουμε απ' όλα. Έχει σημειωθεί ένα σημαντικό άλμα. Τους τελευταίους μήνες ένα 25% του συνολικού διαθέσιμου ποσού. Το 1 τέταρτο θα έλεγα και αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάει σε ένα ποσοστό επιλογής από 25% σε 50% του φακέλου. Βεβαίως αυτό σημαίνει πως τελικά θα πρέπει να πάμε και σε συγκεκριμένες αιτήσει και πληρωμές. Αλλά η λιγότερο θετική πτυχή σημαίνει πως είμαστε πίσω και από το 2007-2013 που δεν είχε ξεκινήσει και πολύ καλά. Και εδώ πέρα δεν θέλω να σας κρύψω ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία οι πιστώσεις ε, πληρωμών ε, που ήταν διαθέσιμες ε, στο προπολογισμό του 2017 δεν θα χρησιμοποιηθούν λυπηρό, αλλά έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Η διαδικασία λοιπόν να ανακτήσουμε τις καθυστερήσεις ε, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Για τις καινοτόμες δράσεις σε αστικά περιβάλλοντα. Πράγματι έχουμε υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μία πρόταση κανονισμού για την παράταση των καινοτόμων προγραμμάτων στα πλαίσια των αστικών δράσεων, τις οποίες καλούμεθα να επιλέξουμε. Αυτό παραμένει για την επόμενη περίοδο, προγραμματίζεται δηλαδή για τον επόμενο Νοέμβριο ουσιαστικά, είμαστε όμως πεπισμένοι από αυτά τα οποία ακούσαμε μέχρι τώρα σαν αντιδράσεις από τις πόλεις και από τις αστικές περιοχές οι οποίες σημείωσαν επιτυχία ε, στον πρώτο διαγωνισμό και τώρα ολοκληρώνουν τα προγράμματά τους ότι δύο χρόνια είναι πάρα πολύ λίγο, ε, μάλλον αρκετά λίγο, για να μπορέσουν να βγάλουν όλα τα απαιτούμενα συμπεράσματα και την πιθανή επανάληψη ε, των, σε άλλη περιοχή των εμπειριών αυτών. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε μέσα από αυτή την πρόταση της κατεξουσιοδότηση πράξης να περάσουμε σε ε, ένα, θα έλεγα, μέγιστο χρόνο διάρκειας 3 ε, ε, με 4 χρόνια. Για τις δράσεις τώρα επικοινωνίας και πληροφόρησης. Θα μπορούσα να σας ενημερώσω εδώ πιο αναλυτικά. Ενθυμίστε ίσως ότι έχει υπάρξει μια κοινή πρόταση για ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο είναι διοργανικής θα έλεγα φύσεως, εμπλέκει και είναι δεσμευτική και για τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και προτείνεται από τις Επιτρόπους Κρέτσου και Τάισεν τον Ιούνιο του 2017. Από δικής μας πλευράς εμείς έχουμε πιέσει με ένα δικό μας πρόγραμμα. Να αναφέρω εδώ ότι έχουμε προχωρήσει τώρα ιδιαίτερα και στους τέσσερις τομείς παράλληλα. Ο πρώτος τομέας είναι για την εκστρατεία ενημέρωσης προς το κοινό είναι κάτι το θα έλεγα αρκετά κλασικό. Ο τίτλος θα είναι «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει στις περιφέρειες». Βρισκόμαστε στην τελική φάση. Αυτό έρχεται αμέσως μετά από μια συντονισμένη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επενδύσεις οι οποίες έχουν υποστηριχθεί από μέσα ευρωπαϊκά. Περιλαμβάνονται εδώ και ε, προγράμματα στη συνοχή, στα πλαίσια της συνοχής και προγράμματα στα πλαίσια των στρατηγικού ταμείου και είμαστε ευχαριστημένοι ότι ε, τα προγράμματα για τη συνοχή έχουν τύχει μεγάλης θα έλεγα προσοχής στα πλαίσια του λεγόμενου EU Invest. Αν σαν παράδειγμα πάτε στο Φιουμιτσίνο, ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο, θα δείτε ένα τεράστιο πίνακα ε, για το πρόγραμμα αυτό. Είναι πολύ ελκυστικό είναι η άποψή μου το, ο πίνακας αυτό, το ταμπλό αυτό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και αρκετά πιστικό θα έλεγα. Συνεπώς λοιπόν έχουμε πετύχει κάποια σημαντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα εμφανή θα έλεγα, στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας. Αλλά όπως είπα θα υπάρξει μια ειδική ε, προσπάθεια με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσφέρει στις περιφέρειες». Επίσης θα επιλεγούν και πρεσβευτές για την νεότητα, θα ασχοληθούν με συγκεκριμένα προγράμματα και που θα επικοινωνούν κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων. Θα θέλαμε τους επόμενους 6 με 12 μήνες να οργανώσουμε και να προκαλέσουμε μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτών ανάμεσα στους πολίτες για την πολιτική της συνοχής. Έχουμε επιλέξει τους εταίρους μας, είναι το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Κοινοτήτων, γνωρίζετε αυτή την οργάνωση και βασικός στόχος είναι να υπάρξουν 60 τέτοιου είδους διάλογοι με το κοινό για την πολιτική συνοχής τους επόμενους 6 με 12 μήνες. Και θα θέλαμε επίσης να υπάρξουν και εταιρικέ συμφωνίες με συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία θα ενημερώνουν πιο συντονισμένα στον τομέα αυτό. Το λέω αυτό συνειδητοποιώντας και όντας ιδιαίτερα ικανοποιημένος ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα κάποια από τα μέλη ε, είναι ιδιαίτερα δραστήρια σε αυτήν την αποκοινού θα έλεγα κινητοποίηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον για την πολιτική συνοχής. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ήταν σαφής και συγκεκριμένη. Θα κάνουμε έναν πρώτο ε, γύρο των συντονιστών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βανίστελ ο οποίος περισσότερο ίσως από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας ε, είναι πρωτοπόρος σε σχέση με το θέμα της εφιούς ε, εξειδίκευσης. Ευχαριστώ, ας είμαστε σοβαροί. Ε, για συγχαίρω για την ομιλία σας για την κατάσταση της Ένωσης. Ε, θα ελέγξουμε την επόμενη εβδομάδα τη ρητορική του Γιούνκερ αν είναι πραγματικά τόσο καλός ρήρος ο ρήτορος ο εσείς. Ε, σε επίπεδο συνοχής έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές προκλήσεις να πω για την ευφυή e e, λοιπόν εξειδικεύση γνωρίζουμε ότι όταν διαπραγματευθήκαμε ε, για τους κανονισμούς <clears throat> που μας ενδιαφέρουν ήταν ήδη σαφές ότι η κυρία Χούμπνερ όταν ήταν επίτροπος και ο επόμενος προχώρησαν σε μια επανατοποθέτηση της πολιτικής μας στα πλαίσια μιας νέας κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης. Και εδώ έρχεται και το ερώτημά μου. Είναι κάτι το οποίο οτθίγει αν θέλετε την εδαφική διάσταση των κοινοτικών πολιτικών. Από τη μία έχουμε το Horizon 2020 και όλες οι εκτιμήσεις τώρα δείχνουν ότι υπάρχουν ε, περισσότερα αιτήματα για χορηγήσεις και όλο και περισσότεροι φοιτητές και καθηγητές που εργάζονται σε ιδρύματα, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η ανάκαμψη της οικονομίας μένει λίγο πίσω. Λοιπόν, αυτά δείχνουν οι αξιολογήσεις και αναφερθήκατε σε αυτό, αλλά στο σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θέλαμε κάτι περισσότερο έτσι ώστε να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι συνέπειες στο ένα το πλαίσιο. Είναι πραγματικά η πρόταση την οποία κάνετε σαν ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο χωρίς ρόδες. Οι ρόδες βρίσκονται στην αποκοινού, θα έλεγα, ιδιοκτησία της καινοτόμου αυτής διαδικασίας και γι' αυτό ξεκίνησα με την κατάσταση των πραγμάτων της Ένωσης, αυτό που σας είπα στην αρχή με το θέμα της καινοτομίας. Αν πράγματι θέλει κανείς να είναι αποτελεσματικός, μπορεί να πει πολλά καλά για την ευφυή εξειδίκευση, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο να έχει σχέση με την Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο, φοβάμαι ότι υπάρχουν κενά. Θα θέλαμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο προχωράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει κάποια κενά στην αξιολόγηση. Δεύτερον, για την ανακοίνωση, χαίρομαι που το ξεκινήσατε αυτό και που μαζί με την Επιτροπή των Περιφερειών και με την ένωση των, για τις αποκεντρωμένες στα πλαίσια της συνοχής δραστηριότητες είναι μια καλή θα έλεγα ευκαιρία να δείξουμε ε, ποια είναι η αξία των πολιτικών μας. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν βοηθηθεί και γι' αυτό Ε, ξεχνάμε τις λεπτομέρειες και καταγγέλουμε πάρα πολύ εύκολα το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσφέρει αυτά που μπορεί. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε με αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι δίνουμε μια προστιθέμενη αξία και στα πλαίσια του Εράσμου σαν παράδειγμα, να τους ενημερώσουμε γι' αυτό και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το επίπεδο σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Μια τελευταία παρατήρηση μαζί με τον εκπρόσωπο της ομάδας των φιλελευθέρων. Είπατε ότι ας βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι σκέφτονται με τον νέο τρόπο να συμπεριλάβουν τέτοιου είδους νέες πρωτοβουλίες και στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ε, δεν υπάρχουν αρκετά μέσα και αρκετό χρήμα έτσι ώστε να έχουμε μια οικονομία η οποία απλά τυπώνει χρήμα. Δεν έχουμε λοιπόν τα χρήματα. Το εύση έχει ίσως κάποια ρευστότητα, αλλά δεν είναι πολύ συγκεκριμένο. Τώρα διαμορφώνεται, οπότε και σύν της άλλης όταν ε, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες υποδομές παραγωγικές, ε, δεν χρηματοδοτεί το εύση. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε μία πρωτοβουλία και αυτοί που είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βάλουμε στο λεγόμενο fast track. Αν έχουμε ας πούμε 21 δις ε, κατανείμει και οι χώρες που έχουν εξοδέψει το 95% ή το 98% μπορούν να περάσουν στην επόμενη φάση. Ενώ ταυτόχρονα αυτοί οι οποίοι καθυστερούν ε, δεν πρέπει να βοηθηθούν πλέον. Αυτοί λοιπόν που δίνουν το καλό παράδειγμα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα αποτελεσματικό fast track. Merci Σας ευχαριστώ. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών η Έλληνα Τζεντήλια είναι ακόμη εδώ. Η Έλενα, όχι. Η ECR, όχι. Φιλελεύθερη. Ελτεμπορκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Λεμέτρ. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος με την πράξη κατεξοδότηση για την επέκταση των αστικών καινοτόμων δράσεων και την περαιτέρω πορεία της ε, αστικής ατζέντα και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποια συνέχεια με κάποιον τρόπο μετά το 2020 των αστικών καινοτόμων δράσεων με περισσότερα κονδύλια με κοινοτική συμμετοχή. Μετά το δεύτερο, η ανακοίνωση και το έγγραφο εργασίας για την ενίσχυση της κοινοτομίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Το έγγραφο έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή όπου έχουμε ακριβώς περιφερειακές στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση που ε, χαράζονται. Έχουμε λοιπόν νέες ε, έννοιες πολύ επιτυχημένες με ιδιαίτερη εστίαση στην καινοτομία, στις περιφέρειες και να δούμε τι θα γίνει βεβαίως και στην πραγματική οικονομία. Αλλά υπάρχει εδώ πέρα κάτι το πολύ σημαντικό το οποίο δεν ε, το ακούσαμε και ελπίζω να επανέλθει σε αυτό. Ε, οι πρωτοβουλίες οι οποίες Φαίνεται οι οποίες είναι πολύ μεγάλες για να χρηματοδοτηθούν σε διεθνή προγράμματα και πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτές που έχουν ένα κάποιο ενδιάμεσο ε, για το πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να βοηθήσουμε τις επενδύσεις εκεί πέρα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη σχετίζεται με την πρώτη, γιατί υπάρχει τώρα η δυνατότητα το 15% των διαθέσιμων ε, κονδυλίων ε, να ε, μπουν στον κάθε προγραμματικό τομέα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό, θα έπρεπε να είναι υψηλότερο. Μπορείτε να μας πείτε τι θα γίνει μετά το 2020, τι προσδοκίες έχετε και τρίτον και βεβαίως ε, να τονίσω την σημασία των προπαρασκευαστικών δράσεων ε, έτσι ώστε ακριβώς να γίνουν ε, εύκολες οι επενδύσεις στο πρόγραμμα Vanguard σε νέες βιομηχανικές υποδομές. Και ελπίζω έτσι μετά το 2020 να έχουμε και δυνατότητες διαρθρωτικής χρηματοδότησης για αυτό το οποίο πολύ σωστά λέτε στην ανακοίνωσή σας για μια συνεργασία μεταξύ των περιφερειών η οποία θα ενισχυθεί. Εκεί πέρα βρίσκεται η πρόκληση για την Ευρώπη για να συνεργαστούμε και με κλάστερς αλλού στον κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. Εκ μέρους των Πρασίνων, ο κύριος Ροπέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία είπατε σε σχέση με τις νέες ιδέες και την εφαρμογή τους σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Για την στρατηγική αυτή που παρουσιάσατε της έξυπνης χρηματοδότησης που δεν είναι ακόμα τόσο γνωστή. Και βεβαίως ε, θεωρώ ότι χρειάζονται περισσότερες και πιο σαφείς ε, πληροφορίες ε, για να μάθουμε περισσότερα για αυτήν την στρατηγική. Και βεβαίω θα πρέπει να πώς θα ζητηθούν οι πληροφορίες, είτε μιλάμε για πόλεις, ε, δήμους, ε, εθνικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα μοιραζόσασταν μαζί μας αυτές τις ε, πληροφορίες. Υπάρχει επίσης παραδείγματος χάρη η περίπτωση της περιφερειάς μου όπου κλείνει ένα πυρηνικό εργοστάσιο και αυξάνεται η ανεργία. Και δεν γίνεται χρήση της πληροφορικής. Έχουμε λοιπόν τους ειδικού, αλλά θα μπορούσαμε νομίζω να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες που υπάρχουν. Επίσης, αναφέρατε ότι δεν είστε ικανοποιημένοι με την χρήση των διαθέσιμων κοντιλίων Και βεβαίως αντιμετωπίζουμε κάποια προγράμματα τα οποία θα έπρεπε ίσως να ενισχυθούν από την Κομισιόν, γιατί εκεί πέρα ακριβώς πάσχει η οικονομία μας και ιδιαίτερα οι φτωχότερες ε, περιοχές ε, που δεν λαμβάνουν κονδύλια για 3-4 χρόνια και κάθε ο κόσμος ε, τρία-τέσσερα χρόνια χωρίς ε, δουλειά και μετά τα επόμενα τρία χρόνια πρέπει να γίνουν όλα τροχάδιν. Γι' αυτό έχουμε την εντύπωση πως ε, δίνεται η εντύπωση πως η Κομισιόν δεν επιτρέπει τίποτα και μετά τα ζητάει όλα μαζί. Και έτσι βεβαίως πάσχει και η αξιοπιστία της Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα διαμορφώσουμε διαφορετικά το χρηματοδοτικό αυτό πλαίσιο και οπωσδήποτε δεν πρέπει να ξεχνάμε το Brexit και βεβαίως αναμένουμε από την ε, Κομισιόν μια διευκρίνηση για τα ζητήματα αυτά. Η Ρόζα Νταμάτο. Ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή λοιπόν για την παρουσία του. Εγώ θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή στο επίπεδο εφαρμογής αν θέλετε της πολιτικής μας ενδιαφέρει από το 14 μέχρι το 20 και θα ήθελα να ζητήσω ένα σχόλιο για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών στην Ιταλία. Εμείς ε, πήραμε από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού τις προγραμματικές ρυθμίσεις ε, της 30ης Ιουλίου 17 μέχρι το 2020 και τα στοιχεία τα οικονομικά δείχνουν ανισχυτικά. Υπάρχουν 72 δις συνολικά και η επιστροφή έχει δώσει μέχρι τώρα 3,9 δις μόνο. Το ποσοστό των πληρωμών σε σχέση με τις υποχρεώσεις είναι πολύ χαμηλού επίπεδου, μόνο 16,2% και μακράν του μέσου όρου που είναι γύρω στο 25% και ισχύει για την Ιταλία, την Κύπρο και την Μάλτα. Το νησιν 3 εφαρμόζεται εδώ που επιτρέπει ένα χρόνο επιπλέον να υπάρξει ε, στη διοίκηση για να μην φύγουν τα χρήματα. Βλέποντας όμως ότι έχει υπάρξει μια αύξηση τις τελευταίες εβδομάδες του ρυθμού σε σχέση με την κατανάλωση των δαπανών, των πιστώσεων, και αυτό δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κανείς συγκεκριμένα στοιχεία. Η Γενική Διεύθυνση Budget έχει επιβεβαιώσει ότι και στη δική της Γενική Διεύθυνση ότι σε σχέση με τον παλιό προγραμματισμό θα έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική μείωση και πάρα πολλά θα χαθούν από τα προγράμματα τα ειδικά για τη συγκυλία και κάποια άλλα προγράμματα για το φυσικό περιβάλλον και τον τουρισμό εκτός και αν υπάρξει στο τέλος μια διόρθωση σε επίπεδο δημοσιονομικό. Πώς λοιπόν έχει αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις στην κατανάλωση των προγραμμάτων αυτών και σε σχέση με τους λογαριασμούς για το 2016 και 2017, τι σκοπεύετε να κάνετε. Σας ευχαριστώ. Δεν ε, θέλει άλλος κανείς το λόγο από, από τους Ζωζεφ Μοσκού πρώτα και ακόμη ένας ομιλητής και μετά θα πατήσετε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω την ανακοίνωση για την έξυπνη εξειδίκευση που μας έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να χαιρετήσω επίσης το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση την ανακοίνωση του περασμένου Ιουλίου για τις στρατηγικές έξυπνης ειδίκευσης. Το έργο δείχνει πόσο απαραίτητη είναι αυτή η στρατηγική που ενθαρρύνει κάθε περιφέρεια να προκρίνει τα ανταγωνιστικά, τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα προκειμένου να καθορίσει τις επενδυτικές προτεραιότητες, ιδιαίτερα για τις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές και αυτές μπορούν με βάση τις ιδιαιτερότητές τους ε, να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους. Βιοπικιλότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, και έτσι θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο δυναμικό καινοτομία, θέσεων απασχόληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά, κύριε Γενική Διευθυντά, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στη δυσκολία του εντοπισμού αυτών των προτεραιοτήτων στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί ναι, είναι σημαντικό να παροτρύνουμε τις περιφέρειες να συνεργαστούμε μεταξύ τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα προτιμούσα να επισημαίνεται και την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας και σε ευρύτερες ε, γεωγραφικές λεκάνες. Για παράδειγμα, τα, υπερπόντια, τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, είτε στον ελληνικό είτε στον ειδικό ωκεανό, ε, ε, εκεί έχουμε πραγματικά γεωγραφικές λεκάνες ε, με τεράστιο δυναμικό ε, συνεργασίας, ε, που όμως δεν αξιοποιείται θα ήθελα λοιπόν και η διαπεριφερειακή συνεργασία να αναπτυχθεί, πέραν όμως και των ευρωπαϊκών συνόρων, όχι μόνο εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Αρίνο Βάκοφ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ε, Μέτρα, σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε και μας μιλήσατε τόσο απλά και κατανοητά και μάλιστα για τόσο περίπλοκα θέματα και μας βοηθάει αυτό τόσο τρόπος με τον οποίο δώσατε τις εξηγήσεις. Πολλές ερωτήσεις ε, υπευλήθησαν και πολλής λόγος έγινε και γίνεται για την έξυπνη ειδίκευση. Εγώ θα σας δώσω μια άλλη σκοπιά αυτού του θέματος. Οι συζητήσεις για την επικείμενη περίοδο προγραμματισμού είναι αναπόφευκτες και πολλές τοπικές και περιφερειακές αρχές ήδη ερωτώνται τι θα γίνει μετά το 2020 και τι μορφή θα λάβει η πολιτική συνοχής. Ε, έχω λοιπόν και εγώ μερικές απορίες και ελπίζω να απαντήσετε. Ποια είναι η γνώμη σας ως προς τη δυνατότητα οι πόροι, ε, τα κονδύλια από τα πέντε διαρθρωτικά ταμεία να μείνουν στον, στα ταμεία και να μην επιστρέφουν στα κράτη-μέλη αν δεν έχουν ε, χρησιμοποιηθεί. Δεύτερον, πώς αξιολογείται σήμερα, πώς εκτιμάτε μάλλον την ιδέα του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων και για τα πέντε ταμεία. Χάρη ε, απλούστευσης, καλύτερης νομοθεσίας, ιδιαίτερα για την πολιτική συνοχή. Και μάλιστα και πριν από λίγους μήνες είχα τη χαρά και την τιμή να, να ακούσω τις ε, ε, απόψες, αλλά μια και οι εξελίξεις ε, είναι δυναμικές, φαντάζομαι θα έχετε και καινούργια στοιχεία ως προς αυτό. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να θέσω μία ερώτηση στον Γενικό Διευθυντή. Πρώτη παρατήρηση. Όντως, ο ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων είναι χαμηλός και αυτό δημιουργεί πρόβλημα Τη στιγμή που προβληματιζόμαστε και πάλι για την περιφερειακή πολιτική ε, με τις πολλές αβεβαιότητες ε, για την περίοδο μετά το 2020. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα και γενικού κλίματος που επικρατεί, αλλά και ως προς το περιεχόμενο. Ε, δεύτερον, φαίνεται ότι δεν μαθαίνουμε πάντα από τα διδάγματα του παρελθόντος. Είμαι και μέλος τη Επιτροπής Προϋπολογισμών και στον προϋπολογισμό του 2018 έχω μια συρρήκνωση των κονδύλιων, αλλά δυστυχώς δεν προβλέπουμε, δεν προλαμβάνουμε ε, τα προβλήματα, γιατί και λόγω αυτής της συρρήκνωσης και της διαφοράς μεταξύ πληρωμών και ανάλυση υποχρεώσεων, πάλι στο μέλλον θα κατακλειστούμε από αιτήσεις για πληρωμές. Γιατί λοιπόν δεν βρίσκουμε πιο βιώσιμες λύσεις, γιατί δεν ε, δασκόμαστε από τα παθήματα του παρελθόντος. Και τρίτον, σε ό,τι αφορά το 2018, μετά από όλα αυτά που σας παρουσίασα, έχετε κάποιες ανησυχίες ως προς την ε, ε, αυτόματη απελευθέρωση. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει σημαντικό τέτοιο ποσοστό αυτόματης απελευθέρωσης ε, κονδυλίων. Αυτά. Ξέρω ότι είναι πληθώρα των ερωτήσεων και ο χρόνος για τις απαντήσεις λίγος, αλλά θα κάνετε ό,τι μπορείτε φαντάζομαι. Ευχαριστώ. Αγαπητά μέλη, Σας έχουν παρουσιαστεί πάρα πολλές και διαφορετικές, κατατεθεί διαφορετικές ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα έγκυρες θα έλεγα, σχετικές και ανήκουν σε μια σειρά δύσκολων ερωτημάτων σήμερα. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι έθεσε ένα δύσκολο ερώτημα όταν συνέκρινε το Horizon 2020 και τις πολιτικές συνοχής, όταν τις ε, έβαλε σε αντιπαραβολή αν θέλετε. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν ε, εύκολο και ε, πολλά υποσχόμενο ε, θα έλεγα δρόμο. Εγώ προήλθα έχοντας παρουσιάσει αυτή την πρόταση σε ένα δείπνο εργασίας για την ανταγωνιστικότητα. Αυτή είναι πολύ πιο κοντά στο Horizon 2020 από ότι εμείς. Εξεπλάγει λοιπόν όταν είδα το τι ακριβώς συμβαίνει στα κράτη-μέλη τους. αναγνώρισα πλήρως αυτού του είδους τις προσπάθειες εκ των κάτω, δηλαδή από τους επιχειρηματίες, από αυτούς προς τα πάνω, οι οποίοι αναγνωρίζουν τις δυσκολίες και οι οποίοι θα πρέπει να συνδεθούν με τη διαδικασία αυτή κάτι το οποίο ενισχύει αν θέλετε τις στρατηγικές μας είναι αυτές οι οποίες θα εξυγχρονίσουν την ε, οικονομία και αν δεν το κάνουμε αυτό νομίζω ότι θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι και θα πληρώσουμε το κόστος. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ανάγκη για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά από τα κάτω προς τα πάνω, ιδιαίτερα για την εφαρμογή της τεχνολογίας. Αναφερθήκατε στην πρωτοβουλία Van Gogh. Συγγνώμη. Στην τροπολογία, στην πρωτοβουλία Van Gogh και στην προσπάθεια δημιουργίας ενός προγράμματος ε, επίδειξης ε, γύρω από την τεχνολογία ε, της, της, τη διάστατη η οποία παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν είναι κάτι που αφορά ένα συγκεκριμένο σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Και υπάρχουν κάποιοι κάποιες βαθιές αλλαγές για την ανανέωση πλέον ορισμένων τομέων μέσω των νέων τεχνολογιών και εκεί ακριβώς η ευφυής e εξειδίκευση μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να ενσωματώσουμε τις προτάσεις αυτές στις ε, παραγωγικές διαδικασίες. Σαν παράδειγμα, υποδήματα πριν 10 χρόνια ήταν κάτι το οποίο θεωρείται στην Ευρώπη ότι ξεψυχούσε. Γιατί, γιατί υπήρξαν ε, βιετναμέζικα, κινέζικα υποδήματα και τι είχε γίνει με τον παραδοσιακό τομέα στις μάρκες της Ιταλία που ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγέας υποδημάτων στην Ευρώπη και για την Ευρώπη ε, για δεκαετίες πριν υπάρξει η λεγόμενη ασιατική εισβολή και επίσης και στο νόρτε της Πορτογαλίας. Και οι δύο αυτές περιφέρειες σε σχέση με την υποδηματοποιία πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Γιατί πηγαίνουν καλύτερα. Γιατί έχουν εν μέρη τουλάχιστον επανεφεύρει ε, τις προσπάθειές τους, ε, έχουν ανεβάσει το επίπεδό τους και έχουν ε, ε, διαμορφώσει και την χρήση τεχνολογιών εντελώς καινοτόμων ε, που ε, προκαλούν ρήξεις με την παραγωγή του παρελθόντος, μεταξύ των οποίων και τους τρισδιάστατους εκτυπωτές. Δεν θα πρέπει εμείς να σβήνουμε λοιπόν τους παραδοσιακούς τομείς και να θεωρούμε ότι θα πρέπει όλοι να γίνουν ειδικοί στις βιοεπιστήμες και την βιομηχανική. Συνεπώς λοιπόν η ευφυής εξειδίκευση εκ των κάτω προς τα πάνω είναι κάτι το οποίο μπορεί να προσφέρει πολλά έτσι ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να πετύχει όσο μπορεί περισσότερα για τις καινοτομίες. Εδώ μπορεί να βοηθήσει το Horizon 2020 και το λέω, μάλλον δεν μπορεί να το κάνει αυτό εύκολα το Horizon 2020 το Horizon 2020 δεν έχει, αν θέλετε, σαν βασικό στόχο αυτό. Όμως εγώ πιστεύω στην ανάγκη και ενός πλαισίου ερευνητικού ε, στην Ευρώπη εκ των άνω προς τα κάτω. Ο όρος τον οποίο εγώ ε, μόνιμα υπογραμμίζω είναι ο όρος συμπληρωματικότητα. Χρειαζόμαστε και τα δύο στην Ευρώπη και δεν θα ήθελα τώρα να μπω σε ένα παιχνίδι αντιπαραθέσεων ανάμεσά τους. Μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία απαιτεί και τις δύο αυτού του τύπου, αν θέλετε, ε, προσπάθειες λογικές και από κάτω προς τα πάνω αλλά και από πάνω προς τα κάτω. Για το Vanguard ε, θυμηθείτε ότι είχαμε πρώτα προτείναμε μια προπαρασκευαστική δράση έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι στόχοι του προγράμματος. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος που βαθμολογείται. Το Β, αν πάρει κανείς Β είναι το χειρότερο, δηλαδή τι γίνεται. Α, όχι, είναι αμέσως μετά από το ε, εξαιρετικό. Θα το κοιτάξω. Ας ε, μου επιτρέψετε τώρα να πω δύο πράγματα γύρω από αυτό. Το πρώτο είναι ότι εδώ έχουμε ένα κενό θα έλεγα στα μέσα μας και πρέπει να καλύψουμε το κενό αυτό στο μέλλον. Αυτό είναι σαφές. Βλέπω δύο τρόπους για να το πετύχουμε αυτό σήμερα και οι δύο ε, αναφέρθησαν και από τον κύριο Μίλτεμπεργκ. Πρώτος είναι να ακολουθήσουμε τη λογική ETC, δηλαδή να έχουμε κάποια διαθέσιμα μέσα σε κεντρικό επίπεδο, μετά η Επιτροπή να κάνει κάποιες προκηρύξεις με κάποιες προϋποθέσεις, περιφέρειες κτλ και στο τέλος να υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση. Είναι απλό και ελκυστικό θα έλεγα το μέσο αυτό. Το δεύτερο θα είναι να το αφήσουμε έτσι, με αποκεντρωμένο τρόπο, στους διάφορους ενδιαφερομένους και να αφήσουμε τελικά την δυνατότητα χρήσης των πιστώσεων που είναι διαθέσιμα ακριβώς μέσα από τα λιταρκικά προγράμματα να λειτουργήσουν σε τοπικό επίπεδο. Προσπαθούμε να δούμε τι επιλογές έχουμε για το μέλλον. Και η δεύτερη παρατήρησή μου εδώ αφορά το εδώ και τώρα. Σε σχέση με το εδώ και τώρα λοιπόν, Έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία τριμερούς διαλόγου για τις προτάσεις Omnibus. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ε, καταθέσει προτάσεις για την τροποποίηση του άρθρου 17. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για το Όμνιμπους και είναι κάτι πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε αν είναι η κατάλληλη στιγμή έτσι ώστε να χαλαρώσουμε τους περιορισμούς και τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στην παρούσα φάση για την χρήση τμήματος των επιχειρησιακών προγραμμάτων για δαπάνες εκτός της γεωγραφικής ζώνης. Απλά το αναφέρω λοιπόν αυτό σαν δυνατότητα. Είναι κάτι το οποίο αξίζει νομίζω τον κόσμο να το σκεφτούμε. Το θέμα σήμερα δεν είναι το 15% γιατί έτσι και αλλιώ οι περιφέρειες έχουν χρησιμοποιήσει το 0%. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι περιφέρειες ε, πρέπει να αποκτήσουν εγγυήσει για τη σωστή δαπάνη αν θέλετε των χρημάτων αυτών και αυτό θα πρέπει να γίνει από τρίτους και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως λίγο τρομάζει τις περιφέρειες. Και δεύτερον, νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και σε πολιτικό επίπεδο η προσπάθεια παρουσιάζει δυσκολίες αν κάποιος που παίρνει αποφάσεις σαν διαχειριστική αρχή πρέπει να δικαιολογήσει το ότι κάποια από τα χρήματα πρέπει να πάνε κάπου αλλού, ακόμα και αν πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον της περιφέρειας, είναι δύσκολο πολιτικά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην επιτρέψουμε να υπάρχουν άλοθη για τις περιφέρειες να μην χρησιμοποιήσουν αυτή την δυνατότητα. αναφέρατε και την διάσταση των πόλεων και το μέλλον αυτής της διάστασης, Μίζον ζήτημα και για μας αυτή η αστική διάσταση και συνεχίζουμε να, επενδύουμε, να στο αστικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εφαρμογή του και οπωσδήποτε θα πρέπει να εγγύψουμε ενδελεχώς αυτό το θέμα και να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε την προσέγγιση του άρθρου 7 με 5% τουλάχιστον προσημείωση και θα πρέπει να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το θέμα που σίγουρα μας είναι προσφυλές και θέλουμε οπωσδήποτε να ενισχύσουμε τις εξουσίες των πόλεων στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Κύριε Ροπέ, για τις στρατηγικές ε, έξυπνης ε, ειδίκευσης ε, διαρωτηθήκατε αν ήταν γνωστές στο κοινό. Ελπίζω, ελπίζω να είναι γνωστές αυτές οι στρατηγικές, αλλά εξαρτάται φυσικά σε ποιο επίπεδο έχει αναπτυχθεί κάποια στρατηγική. Αν δεν κάνω λάθος για τη Λιθουανία τουλάχιστον, έχουμε μόνο μία εθνική στρατηγική. Έξυπνη ειδίκευση. Αν δεν κάνω λάθος, επαναλαμβάνω, αλλά κατά πάσα πιθανότητα έχω δίκιο. Είχαμε δηλαδή μία εθνική διαδικασία στη Λιθουανία. Ε, επιχειρηματιών, ε, επιχειρηματικής ε, αναζήτησης, συμμετοχή του δημόσιου τομέα και της διοίκησης, αλλά και των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων, του ιδιωτικού τομέα και κατά πάσα πιθανότητα και της κοινωνίας των πολιτών. Και αν κάτι τέτοιο γίνεται σε εθνικό επίπεδο, φυσικά δεν έχουν γνώση οι πάντες, ούτε όλοι συμμετέχουν. Αλλά όταν γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και είναι καλά οργανωμένο, και εδώ η διαδικασία έχει μεγάλη σημασία, για να περάσουμε συγκεκριμένα συμφέροντα που θα υπάρχουν, γιατί είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί μια διαφανή διαδικασία, αν όμως είναι καλά οργανωμένη διαδικασία και διαφανής, τότε κανονικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ενημερωθεί λόγω της προπαρασκευαστικής διαδικασίας που προηγείται ε, της έγκρισης της στρατηγικής αυτής της έξυπνης εξειδίκευσης. Οπότε ε, γνωστοποιείτε το θέμα στους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον. Βέβαια, εδώ έχουν ευθύνη οι αρχές διαχείρισης και όχι εμείς. Πρέπει να ξέρουν ότι θα πρέπει να επενδύσουν στην καινοτομία, γιατί αυτό αφορά τη στρατηγική. Και στις ε, προκηρύξεις ε, διαγωνισμών θα πρέπει να υπάρχει σαφής μία αυτής αυτών των στρατηγικών έξυπνης ειδίκευσης όταν ζητούμε και θέλουμε να προσελκύσουμε καινοτόμα σχέδια. Και αυτό είναι ένα άμεσο και φυσικό τρόπο να ενημερωθεί κάποιο για τι στρατηγικέ και το περιεχόμενό του. Προκειμένου να γίνει και αυτό για τους διαχειριστές σχεδίων, το αργότερο σε αυτή τη φάση της προκήρυξης των διαγωνισμών. Μιλήστε για το κλείσιμο ενός πυρηνικού εργοστασίου όντως ε, εύστοχο παράδειγμα και συναφές με αυτά που είπα και εγώ. Θέλουμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και για τέτοιους σκοπούς. Ως σημεία αφετηρίας δηλαδή, μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μια οικονομική μετάβαση και μετασχηματισμό και αναφέρθηκα στις, ε, παραγωγές, στις περιφέρειες ε, που είχαμε παραγωγή άνθρακα και ο αντιπρόεδρος ε, Σεφσοβιτς γνωρίζεται ότι πρόβαλε ιδιαίτερα αυτό το θέμα της οικονομικής μετάβασης ή μετασχηματισμού των ανθρακοπαραγωγών περιφερειών. Αλλά και το δικό σας παράδειγμα ήταν σωστό. Και στην περίπτωση της Λιθουανίας ίσως χρειαστούν περισσότερες τοπικές στρατηγικές, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει, μια και έχουμε μόνο μια εθνική στρατηγική. Πολλές ερωτήσεις ε, στράφηκαν γύρω από το ρυθμό εφαρμογής και ο κύριος Βανίστερο το έθιξε. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε, τι μέλη γενέστε, ε, αν όντω αντλούμε κάποια διδάγματα από το παρελθόν και ούτω καθεξής. Πάντως πιστεύω ότι σήμερα η πιο ενοχλητική διάσταση της ε, παρούσας κατάστασης είναι το γεγονός ότι πλησιάζουμε και μάλιστα ίσως το αναφέρει και στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ο κ. Γιούγκερ πότε θα καταθέσουμε τις προτάσεις για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάντως πλησιάζουμε στην κρίσιμη συζήτηση που θα ξεκινήσει εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάρθρωση του επόμενου, τη δομή του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και την κατανομή των κονδυλίων στους διάφορους μηχανισμούς. Και σίγουρα σε μια τέτοια περίοδο δεν είναι σωστό να δίνουμε την εντύπωση ότι αργοπορούμε. Κάποιοι θα πούν ότι σας έχουν περισσέψει πολλά χρήματα και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι κάτι που με δυσαρεστεί. Είναι και το πιο ενοχλητικό. Πάντως δίκιο έχετε ότι έχουμε εξαγγείλει με ένα πιθανό κύμα ετοιμάτων πληρωμών που θα φτάσει κάποια στιγμή. Πότε? Το 2020, το 2021, 2022, 2023. Όταν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρτίζεται πια από 27 μέλη και όχι 28. Ναι, όντως, μάλλον θα τα βρούμε σκούρα στο μέλλον. Τώρα, με ρωτήσατε, αυτό σημαίνει ότι δεν διδαχθήκαμε από τα παθήματα του παρελθόντος. Ναι, αλλά δεν ήταν ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το, το 3. Δεν ήταν τμήμα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 3 και ξέρουμε που, γιατί καταλήξαμε σε αυτό. Γιατί ακριβώς στην περίοδο εκείνη θέλαμε ένα αργό ρυθμό πληρωμών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήθελε να μην προχωρούν πολύ οι πληρωμές στην περίοδο αυτή. Γι' αυτό πρότεινε το 3. Αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι το παρόν πλαίσιο επιβάλλει μηδενική πειθαρχία. Καμία απολύτως πειθαρχία, γιατί το νησιν 3, ο κανόνας είναι νησιν 3. Αν τα λάβετε όλα μαζί, προκαταβολές και ούτω καθεξής, το νησιν 3 γίνεται νησιν 4 τελικά, ή νησιν 5. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα, σε αυτή την κατάσταση. Γιατί Όλοι έχουμε πείρα από το πώς λειτουργεί ο δημόσιος τομέας. Το δημόσιο είναι εξορισμού βραδικίνητο. Και αυτό είναι ένα μάθημα για το μέλλον και ελπίζω να μην το ξεχάσουμε για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ήδη ξεκάθαρα στο έγγραφο προβληματισμό για τα, το μελλοντικό, με, μελλοντική δημοσιονομική κατάσταση, θέλουμε περισσότερη πειθαρχία στο μέλλον και κάτι παραπάνω. Και αυτό ίσως είναι ένα μάθημα που θα πρέπει να διδαχθούμε από την παρούσα περίοδο και δεν το έχουμε διδαχθεί από τις προηγούμενες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ομαλή μετάβαση από τη μία περίοδο στην άλλη και όχι συνέχεια σταματούμε και αρχίζουμε από την αρχή. Δηλαδή θα, να μην μισολαβούν μεγάλα κενά διαιτίας. Θα πρέπει να έχουμε μια ομαλή εύρυθμη διαδικασία. Έχουμε μια σειρά προγραμμάτων και σχεδίων. Μερικά τα καταφέρουμε να τα χρηματοδοτήσουμε από την προηγούμενη περίοδο και τα υπόλοιπα αμέσως με την έναρξη της επόμενης, χωρίς κενά. Και γι' αυτό δεν πρέπει συνέχεια να τροποποιούμε άρτην το σύστημα. Ναι, μεν θέλουμε απλου, απλούστευση, αλλά να μην επανεφεύρουμε τον τροχό κάθε φορά. Και στις λεπτομέρειες των κανόνων θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να υποφεληθούμε από μια φόρα που έχουμε πάρει ήδη, από μια όθηση προς το από το τέλος μιας περίοδου, ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η φόρα στην αρχή της επόμενης περίοδου. Και αυτό θα είναι πολύ καλύτερο και για την οικονομία να μην υπάρχουν, τέτοιες, να μην υπάρχουν κοιλιές για δύο-τρία χρόνια και δεν κινείται φίλο χωρίς καμία επένδυση. Οπότε στείλαμε το μήνυμα νομίζω ξεκαθαρά για το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης και είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώσουμε την κατάσταση Λοιπόν, για το Brexit, αν κατάλαβα καλά, αναφερθήκατε στα στατιστικά αποτελέσματα του Brexit. Νομίζω πως ε, ήδη είπαμε ότι τα στατιστικά αποτελέσματα του Brexit θα είναι ότι το μέσο ΑΕΠ κατά κεφαλήν ε, της Ένωσης θα μειωθεί κατά 1%. δεν είναι νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό και νομίζω ότι θα πούμε ότι στην έκθεση συνοχής που θα βγει αρχές Οκτωβρίου θα διαβάσετε κάτι σχετικό ούτως ή άλλως θα είναι 300 σελίδες θα έχετε πράγματα να διαβάσετε και νομίζω ότι θα αναφέρετε και αυτό. Κύριε ματο, αυτή τη στιγμή δεν ε, μπορώ να σας δώσω κάποιες ξεκάθαρες πληροφορίες για τη διαδικασία κλεισίματος. Τα κρατη Έχουμε ξεκινήσει, τα κράτη-μέλη έπρεπε να στείλουν τις τελικές εκθέσεις εφαρμογής τον Μάρτιο. Έκτοτε το έχουμε αναλύσει, είχαμε πέντε μήνες. Έχουμε στείλει στην απλούστερη περίπτωση επιστολές κλεισίματος, αλλά δεν είναι πολλές αυτές. Ε, ε, χούφτα ελάχιστες. Και στις υπόλοιπες ζητήσαμε διευκρινήσεις, ε, επιπρόσθετες πληροφορίες κτλ. Εκεί βρισκόμαστε, οπότε φέτος δεν θα κλείσουμε πολλά προγράμματα από το 2007-2013 και πραγματικά αναμένουμε το μεγαλύτερο μέρος να έχει κλείσει το 2018 και το 2019 αρκετά. Να ελπίζουμε το τέλος του 2019 να έχουμε τελειώσει. Ζητήσατε πληροφορίες ε, στα αναδρομικά έργα. Αυτές μπορούμε να σας τις ε, δώσουμε. Βεβαίως ενδιαφέρεστε ε, ειδικά για τις ε, περιφέρειες της Ιταλίας. Ναι, υπήρχαν ε, αρκετές. Γενικότερα θα έλεγα ότι οι παρατηρήσεις σας δείχνουν κάποιες αδυναμίες σε διοικητική ικανότητα και νομίζω ότι μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες για να υπάρξει μια αύξηση ε, των διοικητικών ικανοτήτων μέσω τεχνικής αρρωγής αλλά όπως ξέρετε και μέσω του θεματικού στόχου υπαριθμών 11 και κοιτώντας ε, τα γεγονότα φαίνεται ότι δεν θα έχει τελειώσει η δουλειά μέχρι το τέλος αυτής της ε, περίοδου και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Κύριε Μοσκούρ, το θέμα που θίξατε της ε, συνεργασίας σε ευρύτερες γεωγραφικές λεκάνες θα περιληφθεί στη μελλοντική μας ανακοίνωση για μια ανανεωμένη στρατηγική για τις ε, περιφέρειες και συγκεκριμένα κάνουμε ένα απολογισμό της παρούσας κατάστασης για να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα διάφορα ταμεία και κονδύλια. Τώρα για συγκεκριμένες δυσκολίες. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα την κατάσταση για ένα συγκεκριμένο σχέδιο βιολογικού καθαρισμού στον Άγιο Μαρτίνο, το Σεντ Μάρτιν. Ε, το Ολλανδικό Τμήμα θα πρέπει να παράσχει τη χρηματοδότηση μέσω του ΦΕΤ, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, του ΦΕΔ, μάλλον και το ΣΕΜΑΧΤΑ, το γαλλικό τμήμα μέσω του ΦΕΝΤΕΡ. Διαπιστώνουμε ότι δεν είναι πρόβλημα κανόνων και έχουμε την το πρώτο παράδειγμα τέτοιων ε, μεικτών σχεδίων, κοινών σχεδίων. Αλλά ε, υπάρχει ένα πρόβλημα με έναν εταίρο και μάλιστα που δεν αφορά καν την περιφέρεια, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία μάλλον στο συγκεκριμένο θέμα. Πάντως οι κανονιστικές δυσκολίες και δεν μιλάω για τις πολιτικές. Οι κανονιστικές δυσκολίες αυτών των συνδυασμών είναι, των είναι μεγάλες. Και γι' αυτό θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα πιο εύκολο σύστημα για τέτοια κοινά σχέδια και προγράμματα μεταξύ εδαφών της Ένωσης και τρίτων ε, αλλά περιφερειών ή εδαφών. Πάντως, στην ανακοίνωση ε, για την ανανεωμένη στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές ε, θα αναφέρεται το θέμα αυτό. Την περιμένουμε για τα τέλη Οκτωβρίου, συγγνώμη. Τέλος, ε, κύριε Νοβακόφ, ανακύκλωση των κονδυλίων που έχουν αποδεσμευτεί έχει προτείνει η Κομισιόν σε γενικές γραμμές εντός του Ομνιμπούς να γίνει αυτό. Το Συμβούλιο δεν έχει μεγάλη όρεξη να κάνει κάτι τέτοιο η διαδικασία του τριμερούς διαλόγου εντάξει, μπορεί να το αλλάξει, αλλά αυτή ήταν η αρχική μας πρόταση και βεβαίως ε, το σκεπτικό ήταν να έχουμε ένα γενικό αποθεματικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στον κοινοτικό προπολογισμό και οπωσδήποτε εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι ε, αυτό θα είναι μια σημαντική βελτίωση για την διαχείριση του προπολογισμού. Λοιπόν, ενιαίοι κανόνες. Ε, δείτε και πάλι το έγγραφο που έχουμε κάνει, το έγγραφο σκέψεων, το αναφέρουμε και με τρόπο θετικό νομίζω. Αλλά είναι ένα έγγραφο σκέψεων της Κομισιόν παρόλα αυτά. Δεν είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση της Κομισιόν ακόμα, αλλά εμείς προς τα εκεί θέλουμε να πάμε. Και προς τα εκεί προωθούμε τα πράγματα όσο μπορούμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό για την απλοποίηση. Και αυτό πηγαίνει πέρα από τα κονδύλια του Ταμείου Στρατηγικών Επιμήσεων. περιλαμβάνουμε τους ίδιους κανόνες ε, για τις κρατικές ενισχύσεις και με τα διάφορα μέσα, τον ορίζοντα 2020 και τις δημόσιες προμήθειες. Και επανέρχομαι τέλος στο θέμα της απορρόφησης με δύο λόγια. Μακάρι να υπήρχαν κάποια κίνδυνοι για τις αυτεπάγγελτες ε, απελευθερώσεις. Αυτό θα έδειχνε μια κινητοποίηση των κρατών μελών. Δυστυχώς όμως, αν εξετάσουμε το μηχανισμό του νησιν 3, όπως έχει εφαρμοστεί, δεν μιλάμε ουσιαστικά για νησιν 3, αλλά για νησιν 4, νησιν 5 και το καθεξής. Και δυστυχώς, δυστυχώς δεν υπάρχει καν κίνδυνος για τέτοιες αυτεπάγγελτες αποδεσμεύσεις για το 2018. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν ε, πιέσει στα κράτη-μέλη για να κάνουν σοβαρές επιταχύνσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε ε, Γενική Διευθυντά ήταν πολύ ε, συγκεκριμένη, απτή, δυναμική συζήτηση με μεστή και χάρη σε αυτή διαμορφώσαμε μια πιο ξεκαθαρή άποψη για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούσαν και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν και στο μέλλον. Πάντως ε, ακούσαμε με προσοχή και την αρχική σας παρουσίαση και τις διευκρινήσεις για τις κατεξοδότηση πράξεις και για την εφαρμογή κάποιων καινοτόμων δράσεων στα, στις πόλεις. Μιλήσατε για παράταση της προθεσμίας από 3 4 χρόνια και ε, ξέρω ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολή αντιρρήσεων εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα σε ένα δίμηνο ή αίτηση ε, για περίοδο προβληματισμού, προθεσμία προβληματισμού για ένα επιπλέον δίμηνο. Οι συνάδελφοι έχουν λάβει ε, στοιχεία και πληροφορίες από τη γραμματεία μας και ακούσαμε και τις εξηγήσει ε, του Γενικού Διευθυντού για το θέμα αυτό. Οπότε, με βάση όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε και ακούσαμε το απόγευμα, εγώ θα πρότεινα να μην καταθέσουμε ένσταση, αντίρρηση. Έχει κανεί αντίρρηση για την πρότασή μου να μην υποβάλλουμε αντιρρήσεις ή ενστάσεις. Ωραία, πολύ ωραία. Και σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε σε άλλη ευκαιρία για να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο. Οπότε, σας αφήνω ένα λεπτό για να αποχωρήσετε. Και θα περάσουμε στην γνωμοδότηση του κύριου Χέτμαν, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την υπομονή του. Ε, θα μας παρουσιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, έκθεση και ε, γνωμοδότηση και πολύ σημαντική για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Χέτμαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάστηκε καθόλου υπομονή, επίδειξη υπομονής, γιατί συμφωνώ μαζί σας ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική συζήτηση. Επανέρχομαι στο δικό μου θέμα, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Πρόκειται για τη δεύτερη συζήτηση για το θέμα αυτό και στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε μια αρχική ανταλλαγή απόψεων με βάση το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ενημερωθήκαμε για το έγγραφο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα όλοι γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είχα πει την περασμένη φορά. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα στην διαμόρφωση της γραμματότησης ε, μετά και την υποβολή των τροπολογιών. Δεν θα αναλύσω διεξοδικά τις τροπολογίες, θα σας κάνω μια γενική παρουσίαση της κατάστασης. Καταρχήν, θα ήθελα το σχέδιο γνωμοδότησής μου να έχει πολύ σημαντικό χαρακτήρα και να βάλει το στίγμα το τοπικό και το περιφερειακό, γιατί στα πλαίσια του εθελοντισμού, των πρακτικών ασκήσεων και άλλων απασχολήσεων, θα έχουν την ευκαιρία πολλοί νέοι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να ενταχθούν. Γι' αυτό είναι σημαντικό στο έγγραφό μας να αναγνωρίσουμε τον τοπικό και περιφερειακό χαρακτήρα αυτού του, του σώματος αλληλεγγύης. Και τώρα, στο έγγραφό μου ε, λέμε ότι η ιδέα του σώματος ε, ε, και το πρόγραμμα θα πρέπει να συνάδει με τα εθνικά προγράμματα. Και θα έλεγα να εξασφαλίσουμε συνάφεια και με τα περιφερειακά και τοπικά προγράμματα, όχι μόνο με τα εθνικά. Είναι σημαντικό να δώσουμε το τοπικό και περιφερειακό στίγμα, γιατί σίγουρα όλα αυτά τα προγράμματα εθελοντισμού, πρακτικών ασκήσεων κτλ. πρέπει να εξυπηρετούν τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες. Ένα άλλο σημείο που είχα θίξει και στην προηγούμενη συνεδρίαση κατά την παρουσίαση του σχεδίου, για μένα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Υπήρξε πρόταση για ε, το 80 με 20%, δηλαδή 80% για το εναθελοντισμό και 20% για, την, για το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Είναι ε, λεπτό αυτό το θέμα ε, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντική προστιθέμενη αξία για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση για του νέου αυτό. Ε, πολλά δε μάλλον που η ανεργία των νέων σε πολλέ χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε δραματικά υψηλά επίπεδα. Ε, ιδιαίτερα για του νέου που είναι στο στόχαστρο του σώματος Ελληνική, δηλαδή νέου μέχρι 30 χρονών. Γι' αυτό και προτείνω να αλλάξουμε τα ποσοστά και ο λόγος να έμεινε 80-20 αλλά 70-30, δηλαδή 30% για τις ε, νέες θέσεις ε, απασχόλησης και πρακτικής άσκησης. Επίσης, ε, μιλήσαμε για τα άτομα με αναπηρίες. Ε, μην ξεχνάτε το έγγραφο για την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες. Και εδώ προβλέπεται και κοινωνική βοήθεια στα πλαίσια του σώματος αλληλεγγύης, αλλά ε, κρίνα σωστό στην τροπολογία 5 να αναφέρουμε ρητά ε, τη δραστηριότητα αλληλεγγύης και για τα άτομα με αναπηρίες, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ε, είναι και αυτοί ε, οι άνθρωποι μέσα. Επίσης προτάθηκε η συνεργασία για την υλοποίηση αλληλέγγυων σχεδίων και προγραμμάτων να περιοριστεί σε πέντε εταίρους. Εγώ ε, προτείνω να αναφέρουμε την ε, περιφερειακή διασυνοριακή συνεργασία χωρίς περιορισμό του αριθμού των εταίρων. Δεν βλέπω από πρακτική άποψη προς τι ο περιορισμό. Γιατί θα πρέπει εμείς να καθορίζουμε πόσοι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην υλοποίηση. Μερικέ φορέ μπορεί να χρειάζονται δύο ή τρει. αλλά σε άλλη περίπτωση να χρειάζονται έξι ή εφτά. Γιατί να περιορίσουμε τον αριθμό των εταίρων σε πέντε. Επίση. θα ήθελα να φέρω κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμη στο σχέδιο γνωμοδότησης, αλλά θα ήθελα να το λάβουμε υπόψη στη συνέχεια των εργασιών μας. Και μάλιστα πρόκειται για κάτι που προέκυψε από μία πρακτική και μία κατάσταση που ανέκυψε δυστυχώς το τελευταίο 1,5 μήνα. Ε, το σεισμό στην Κόενο Ήταν τραγικός και ο σεισμός γιατί είχαμε ανθρώπινα θύματα, αλλά και το τελευταίο ε, μήνα είχαμε τραγικά προβλήματα στην Πολωνία στο βόρειο τμήμα. Ε, μάλιστα αυτό το εργαλείο ίσχυε από τον ε, Ιούνιο και ε, σκέφτηκα να το αξιοποιήσω, να αξιοποιήσω αυτό το μηχανισμό και να επιστήσω την προσοχή των ενδιαφερόμενων τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Πολωνία και την Ελλάδα και να τους επισημάνω ε, τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν εθελοντέ στα πλαίσια αυτή τη της για το σώμα αλληλεγγύη, ιδιαίτερα σε τέτοιες περιπτώσεις ε, ε, θεομηνιών. Και φαίνεται ότι το σημερινό σύστημα που λειτουργεί θα οδηγούσε οι πρώτοι εθελοντές να φτάσουν στο, στις πληγείς περιοχές το νωρίτερο του χρόνου το Φεβρουάριο. Γι' αυτό και κατέθεσα σχετική τροπολογία για να επισπευστεί αυτή η προθεσμία, γιατί κατόπιν ορτής ε, δεν εξυπηρετεί αυτή η βοήθεια ούτε για, το, για τους τοπικές κοινότητες, ούτε για τους αναπήρους και ενώ μερικές φορές οι τοπικές κοινότητες ή οι ανάπηροι μπορούν να περιμένουν να διεκπαιρεωθεί η διαδικασία, στην περίπτωση θεομηνίας έχει σημαντικό χαρακτήρα η αμεσότητα της βοήθειας. Θα πρέπει οι εθελοντές να μπορούν άμεσα να μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές. Τότε είναι που χρειάζονται οι σεισμόπληκτοι, οι πλημμυροπαθείς ή τα θύματα οποιασδήποτε θεομηνία στη βοήθεια από τους εθελοντές. Γι' αυτό, στη γνωμοδότησή μου, ε, θα αναφερθώ στη διαδικασία άμεσης αξιοποίησης των εθελοντών για να μην υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις. Καλό θα ήταν αυτό το θέμα να το λάβουν υπόψη ε, οι συντάκτες ε, των προτάσεων για το Σώμα Αλληλεγγύης. Αυτά από μένα. Περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων για μια διεξοδική ελπίζω συζήτηση και φυσικά περιμένω και τις υπόλοιπε τροπολογίες σας. Και παραλαμβάνω αυτό που είπα και στην πρώτη σα Συγχαρητήρια ε, στην Επιτροπή για το πολύ αξιόλογο έγγραφο που εκπώνησε. Γιατί ήταν τόσο άρτιο το έγγραφο που ήταν δύσκολο ακόμη και τροπολογίες να καταθέσουμε, γιατί ήταν ελάχιστα τα σημεία που ε, υπήρχαν κενά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσίασή σας. Θα πρέπει να πω ότι με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει πραγματικά να αγαπηθεί από τους πολίτες. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι επί της ουσίας υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Πολιτισμού και στην πρόταση του συναδέλφου τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για το ότι επιμένει στις τοπικές κοινότητες και στην περιφερειακή διάσταση. Είναι μια προστιθέμενη αξία, αν θέλετε, σχετικά με την αρχική πρόταση της Επιτροπής Πολιτισμού. Η κυρία Τζεντήλε, η συγγήτρια Σκιώδης για τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα το οποίο είναι η υποσυζήτηση εδώ νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. γιατί μας δίνει την δυνατότητα να εφαρμόσουμε με συγκεκριμένο τρόπο την επικουρικότητα, την αμοιβαία αναγνώριση των διαφορών ιδιαίτερα σε μια χρονική στιγμή όπου δυστυχώς οι εθνικιστικές τάσεις προσελκύουν ε, πολλούς νέους που θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν είναι μια μεγάλη ευκαιρία αλλά ένα απλό ατύχημα ιστορικό. Το μέσο αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για όλους μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε τις τάσεις αυτές. Και εμείς σαν κοινοβούλιο που είμαστε φίλο Ευρωπαίοι θέλουμε να επιβάλλουμε τις ε, πολιτικές μας επιλογές. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι έτσι κι αλλιώς το μέσο είναι έγκυρο, είναι χρήσιμο και στο μέλλον θα είναι και αποτελεσματικό. Να υπογραμμίσω όμως την ανάγκη η οποία υπάρχει να καθορίσουμε ε, με συγκεκριμένο τρόπο το τι είναι η εθελοντική προσφορά και το τι μας προσφέρει μια ανάγνωση, αν θέλετε, ε, σε διαφορετικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει αντιφάσεις, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε έλλειψη ισορροπίας αυτό που μας ενδιαφέρει. Αυτοί οι οποίοι θα θεωρήσουν ότι αυτή η δωρεάν προσφορά σε ένα πρώτο επίπεδο ε, είναι κάτι το οποίο χρήζει εξέτασης, είναι κάτι το οποίο απαιτεί μια κλίδα ανάγνωσης με διαφορετικό τρόπο στον χώρο της εργασίας. Η καθαρή εθελοντική προσφορά, αν θέλετε, δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό ασυμβατικό, δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό οικονομικό και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ξεχωρίσουμε καλά τα δύο πράγματα. Αυτά θα πρέπει να καθοριστούν σωστά λοιπόν, όπως θα πρέπει να καθοριστούν σωστά και οι ευθύνες τις οποίες έχουν τα κράτη-μέλη. Το θέμα εδώ είναι πάρα πολύ περίπλοκο και γι' αυτό θα ήταν χρήσιμο, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, να υπογραμμίσουμε το θέμα του καθορισμού των ευθυνών σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο τοπικών αρχών. Γιατί νομίζω ότι στο εσωτερικό του συστήματος υπάρχουν χώροι για σωστή ενημέρωση σχετικά με τα κατεπήγοντα θέματα έτσι ώστε οι νέοι να είναι σε θέση να επιλέξουν ε, ανάμεσα σε διαφορετικές δραστηριότητες στον περιβαλλοντικό τομέα ή στον τομέα της φροντίδας αυτών που έχουν ανάγκη. Ένα σύστημα δηλαδή το οποίο πρέπει να μπορέσει αντικειμενικά να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα των πόρων που μπορεί να έχει, που πρέπει να έχει αυτή η προσπάθεια, πόροι οι οποίοι σίγουρα θα επηρεαστούν και από εμά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν απορίες λοιπόν, υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις, ιδιαίτερα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές οι οποίες βλέπουν ε, ο προϋπολογισμός τους να αποκεφαλίζεται σε εισαγωγικά, εν μέρη τουλάχιστον. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι εμείς ε, θέλουμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση, αλλά δεν μπορούμε να αποκρύψουμε κάποιες ε, φάσεις οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρες. Σας ευχαριστώ πολύ ε, για τους συντηρητικούς. Κύριε Σκοζουάφσκι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Χέτμαν για την παρουσίαση του σχέδιου γνωμοδότησή του και επίση να τον ευχαριστήσω για τις ενδιαφέρουσε και εύστοχε ε, τροπολογίες του ε, που πλαισιώνουν πολύ καλά αυτό το ενδιαφέρον πρόγραμμα. Γι' αυτό και συμφωνώ και με τις τροπολογίες συμφωνώ ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα αποτελέσει ευκαιρία για την κινητοποίηση πολλών νέων. Και ε, θα δώσει έμφαση σε αυτή την ε, εθελοντική εργασία και τις πρακτικές ασκήσεις, φέροντας στο φως το πόσο σημαντική είναι η Ελληνική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχει και πολύ θετικές ε, δράσεις. Έλειπε κάτι τέτοιο Επίσης, ε, να μην ξεχάσουμε τους πιο ευάλωτους νέους ε, που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και επίσης ε, να λάβουμε υπόψη και τους ανάπηρους νέους γιατί μερικές φορές το κυρίως έγγραφο τους ξεχνά ή δεν δίνει τη προσοχή και στους ανάπηρους νέους και στους πιο ευάλωτους ή τους κοινωνικά περιθωριοποιημένους. Είναι σημαντικό να τους αναδείξουμε ε, και να τους φέρουμε στο επίκεντρο της προσοχής. Επίσης, ε, ε, είναι σημαντικό να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να κινητοποιήσουμε τους νέους σε τέτοιες κοινωνικές δράσεις και σε περίπτωση θεομηνιών. Και είναι επίκαιρη στιγμή μετά αυτά που συμβαίνουν με τον τυφώνα στην Καραϊβική και βλέπουμε πόσο δραματικές είναι οι στιγμές και πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη ε, κινητοποίησης των νέων σε τέτοιου είδους εθελοντικές ε, δραστηριότητες ε, γιατί είναι σημαντικό να μάθουν οι νέοι την κοινωνική ευαισθησία με τη συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις γιατί αυτό έλειπε μέχρι στιγμής. βέβαια το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης χρήζει κάποιων συμπληρώσεων και κάποιων προσθήκων που ελπίζω να γίνουν χάρη και στις δικές μας τροπολογίες, γιατί και ο, ο συντάκτης γνωμοδότησης ήδη ανέφερε και περιέγραψε κάποιες τροπολογίες. Στη συνέχεια θα συμπληρώσουμε τη γνωμοδότηση και με δικές μας. Πάντως, εκ πρώτης όψεως, πιστεύω θα, ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε τις αρμοδιότητες, γιατί ίσως δημιουργήσει κάποια σύγχυση, κάποια προβλήματα στην φάση της εφαρμογής ή τη στρατηγική θέσπιση προγραμμάτων και την συμπληρωματικότητα που θα πρέπει να ισχύει για να μην λειτουργεί αυτό το σώμα αλληλεγγύης εν και ενώ σε σχέση με το, Ευρωπαϊκό, το πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Εθελοντισμού ή το πρόγραμμα Ερασμοσύν. Να μην υπάρχει επικάλυψη. Επίσης, να μην γίνει απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα περισσότερο για αύξηση πρακτικών ασκήσεων ή θέσεων απασχόλησης. Πιστεύω λοιπόν ότι δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες για την ενεργοποίηση των νέων αυτό το σώμα αλληλεγγύης, αλλά ίσως πιο αποτελεσματικός τρόπος στήριξη των νέων και καταπολέμηση της ενεργείας των νέων δεν θα ήταν η ενίσχυση. Ε, μήπως θα ήταν η χρηματοδοτική ενίσχυση των κρατών μελών γιατί τα κράτη-μέλη είναι στην καλύτερη δυνατή θέση να γνωρίζουν τα προβλήματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων τους ή του κοινωνικού αποκλεισμού που μερικές φορές τους απειλεί. Θα πρέπει λοιπόν να σταθμίσουμε και αυτό το θέμα και να το εξετάσουμε. Μήπως όλες αυτές τις δυνατότητες που προσπαθεί να αξιοποιήσει το, σώμα, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα μπορούσαμε να τις καλύψουμε καλύτερα με την οικονομική ενίσχυση των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα των φιλελευθέρων, ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρά το ότι είμαι ένα πληρωματικό μέλος της Επιτροπής, Είναι αυτή τη στιγμή σκιώδης ε, αναπληρωτής για, σκιώδης εισηγητής για αυτό το θέμα και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθεί ένα αίσθημα του ανήκειν ε, για τους ε, νέους ε. για να υπάρξει μια αισθησή ευθύνη σε δραστηριότητες όπου θα εκφραστεί αυτή η αλληλεγγύη. Πρέπει οι νέοι να έχουν την δυνατότητα να βρουν ακριβώς αυτήν την ευθύνη για την κοινωνία γιατί η ευημερία δεν δημιουργείται μόνο από τις αρχές όλοι οι πολίτες ε, θα πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι είναι υπεύθυνοι για την ζωή τους και τη ζωή των άλλων πρέπει να είναι να συνεισφέρουν και να μπορούν να κάνουν κάτι το συγκεκριμένο. Γιατί μόνο οι πράξεις ε, έχουν νόημα. και θα πρέπει οι νέοι, οι νεαροί ενήλικοι να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν. Ειδικά τώρα απαιτείται να υπάρχει δυνατότητα της συνεργασίας. Έχουμε όλα αυτά τα νέα ΜΜΕ, τις ε, ηλεκτρονικές ε, μεθόδους ε, και έχει μεγάλη σημασία πλέον η εμπειρία, η αυτοπρόσωπη κάποιου. Και έτσι νέοι θα αυξήσουν ε, και την υπευθυνότητά τους και αυτό το απλοποιήσαμε ήδη. Αυτό μπορεί να έχει μεγάλη σημασία το μέσο αυτό. Από την τοπική και περιφερειακή πτυχή και πρέπει να ενισχύσουμε αυτήν την ε, πτυχή Ευχαριστώ τον κύριο Χέτμαν για την καλή συνεργασία και θεωρώ ότι μπορούμε έτσι να βελτιώσουμε περαιτέρω την έκθεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι κύριε Χέτμαν, είναι κάτω πολύ θετικό, μια πολύ θετική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πρακτικά νομίζω θα δημιουργήσει μια θετική προσθέμενη αξία για τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι απούσα η εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ για τους πρασίνους τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Χέντμαν για την δουλειά του και εξ ονόματος ε, της ε, συναδέλφου ζητώ συγγνώμη γιατί ψιάζει. Να αναφέρω τα σχόλια των Πρασίνων. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αυτή για να συγκεντρώνουν οι νέοι εμπειρίες ε, που θα τους φανούν χρήσιμες μετά στην αγορά εργασίας και βεβαίως αυτονόητο είναι ότι χαιρετίζουμε την ίδρυση αυτού του σώματος και ειδικά το κομμάτι που αφορά την απασχόληση. κομισιών θέλει να προωθήσει την ε, απασχόληση των νέων. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεγάλη ανεργία των νέων, αλλά ταυτόχρονα δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό μέσο για μείωση της ανεργίας. Ανησυχούμε δηλαδή για το ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πηγή φτηνού εργατικού δυναμικού. Το Erasmus Plus, η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία θα μπορούσαν να κάνουν την ίδια δουλειά. Και δεν θέμε να είναι ανταγωνιστική η μία δομή της άλλης. Πρέπει να επιδιώξουμε την συνέργεια. νομίζω ότι θα μπορούσε έτσι να παίξει μεγάλο ρόλο η δραστηριότητα του σώματος αυτού, τα προγράμματα αυτά μπορούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τις ε, επιτόπιες ε, κοινότητες. Θα πρέπει λοιπόν να εξαντλήσουμε το δυναμικό αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε και το τι θα γίνει με την υλοποίηση κοινωνικών ε, αναγκών επιτόπου. Σας ευχαριστώ η κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα του κύριου Χέτμαν είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγω και των φυσικών καταστροφών τις οποίες παρακολουθήσαμε τα τελευταίο χρόνο και έχει και ιδιαίτερα συμβολική αξία γενικά για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γιούνκερ το 2017 στις αρχές για την κατάσταση της Ένωσης είπε ότι στόχος του σώματος αυτού είναι να δώσει τη δυνατότητα στους νέους να πάρουν μέρος σε αλληλέγγυες δράσεις κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο στους νέους αλλά άπτεται και των προσπαθειών των τοπικών αρχών όπως επίσης και των ΜΚΟ να αντιμετωπίσουν κρίσεις και προκλήσεις. Εγώ είχα ήδη υπογραμμίσει στο παρελθόν ότι έχουμε φυσικά σύμφωνη γνώμη, αλλά έχουμε και κάποιες απορίες για τον προϋπολογισμό. Τα 340 εκατομμύρια για να κινητοποιήσουμε 100.000 νέους, ε, παίρνοντας χρήματα από άλλα προγράμματα όμως. 25 εκατομμύρια, 120 εκατομμύρια από το Erasmus Plus, 10 εκατομμύρια από το κοινωνικά ταμεία κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να αξιολογήσουμε αν υπάρχει δυνατότητα να αυξήσουμε τα 86 εκατομμύρια του μη αναγνωρισμένου πλεονάσματος στο πρώτο τμήμα του προϋπολογισμού γύρω από αυτό προγράμματα αυτά θα συμφωνήσω με την ανάγκη εξισορρόπησης από τη μία της αξιολόγησης του προγράμματος με ένα μηχανισμό ο οποίος να μην κοστίζει ιδιαίτερα σε επίπεδο γραφειοκρατίας επίσης. Να επαναλάβω εδώ τα αποφάσεις που έχει ήδη εγκρίνει το Κοινοβούλιο τον προηγούμενο Απρίλιο και στα πλαίσια των οποίων καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να κάνει μια σαφέστατη διάτρηση ανάμεσα στην εθελοντική εργασία και στην πραγματική αμοιβόμενη εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε προσεκτικά τον τρόπο εργασίας, το περιβάλλον εργασίας, και ε, τις διαφορετικές φύσεις απασχόλησης ε, των εργαζομένων από τη μία στο σώμα και των εθελοντών από την άλλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χέτνερ, έχουμε τον εκπρόσωπο της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο κύριος Φράνς είναι εδώ. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σα Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ και που ε, έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για την πολύ θετική αυτή πρόταση που έχουμε μπροστά μας γιατί με την ε, πρόταση αυτή ε, σκοπεύουμε να δεσμευτούν περισσότερο οι νέοι προς την Ευρώπη και να έχουν περισσότερες ευκαιρίες και θέλω να το πω αυτό για όλους τους νέους. Ε, προσέχουμε λοιπόν να υπάρχει συμπερίληψη όχι μόνο από πλευράς αναπηρίας αλλά για οποιοδήποτε πιθανό και πιθανό εμπόδιο που μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς στην συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια αυτά τα οποία σημειώνουμε και πριν αντιδράσω. Συγκεκριμένα θα ήθελα να τονίσω ακριβώ ε, την ε, σημασία που έχει αυτό στην εφαρμογή του, αλλά βεβαίως και στην διάδοση των πληροφοριών που θα και για τις ευκαιρίες που θα παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Τώρα να περάσουμε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Το ποσοστό αυτό 80-20 μεταξύ εθελοντισμού και εργασίας. Η πρόταση αυτή βασίζεται στον υφιστάμενο προϋπολογισμό με στόχο να μην μειωθούν οι δυνατότητες εθελοντισμού που υπάρχουν στο Erasmus Plus. Ίσως γνωρίζετε ότι το Erasmus Plus στηρίζει αυτή τη στιγμή τις εθελοντικές ε, δραστηριότητες. Για να μην έχουμε λοιπόν και τις δύο δραστηριότητες, ε, τα λεφτά μαζί με τις δραστηριότητες του Erasmus Plus μεταφέρονται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και μιλήσαμε για την συμπερίληψη, οπότε έχουμε προσθέσει κάποιες επιπλέον μορφές, όπως ομαδικές δραστηριότητες ή ε, έργα αλληλεγγύης, οπότε αυτό το 80-20 αντικατοπτρίζει την κατάσταση, ότι δηλαδή δεν θέλουμε να μειώσουμε τις ήδη προτινόμενες θελοντικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τα έργα αλληλεγγύης. Εδώ έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα όπου πηγαίνουμε κοντά στην βάση. Είναι τοπικές πρωτοβουλίες ε, ομάδων νεαρών. Δεν χρειάζεται καν να είναι κάποια οργάνωση. Συνήθω είναι μια άτυπη ομάδα και δίνουμε κάποια χρηματοδότηση μικρή, 5.000 ευρώ και μπορούμε έτσι να φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο τοπικό επίπεδο. Οπότε προτείνουμε να διατηρηθεί στο τοπικό επίπεδο και να μην υπάρξει κάποιο επιπλέον στρώμα και κάποια διεθνής ε, ε, διάσταση. Τώρα να αναφερθώ λίγο στις τεχνικές εκφράσεις ε, του προπολογισμού ε, σημειώνω ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που ζητούν να ξεκαθαρίσουν οι πηγές ε, του βασικού ε, ποσού αναφοράς. Έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα Erasmus Plus, το πρόγραμμα Easy και από το γενικό αδιάθετο υπόλοιπο. Αλλά να εξηγήσω την διαφορά. Αυτή τη στιγμή στον κανονισμό γιατί από τη στιγμή που θα τεθεί ενισχύ ο οργανισμός. Ε, τα ποσά αυτά δεν σχετίζονται πλέον με τις πηγές ε, των προγραμμάτων, αν είναι δηλαδή Erasmus Plus, Easy ή από κάπου Αντιθέτως, σε αντίθεση δηλαδή με τα κονδύλια των ταμείων που αναφέρονται παρακάτω, όπως το πρόγραμμα Life. Και αυτό οφείλεται στο ότι το δεύτερο αυτό ποσό παραμένει στους τίτλους όπου αρχικά ήταν και θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τους στόχους των προγραμμάτων αυτών. Οπότε υπάρχει μια διάκριση που πρέπει να γίνει. Αντιλαμβάνομαι την πολιτική ανάγκη ε, για να ξέρετε από πού προερχόνται τα λεφτά. Αλλά θα δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν να εκφραστεί κάτι τέτοιο στον κανονισμό. Επίσης σημειώνω το ότι υπάρχει μια πρόταση να συλλέγονται εκθέσεις συμμετεχόντων. Είναι μια πρακτική που έχουμε ήδη στο Erasmus Plus, στην εθελοντική υπηρεσία. Για εμένα, δεν ξέρω, εξαρτάται το ε, εάν ε, η ρητή αναφορά τέτοιου πράγματος στον ε, κανονισμό που κάνει ε, την κατάσταση πολύ δύσκολη. Π.χ. κάποιοι διακόπτουν την υπηρεσία του λόγω, για λόγου υγεία ε, κάποιον τραυματισμό. Ε, δεν ξέρω αν χρειάζεται όλοι αυτοί να υποβάλουν αναφορά. Τέλος, δύο πράγματα ακόμα. Το ένα είναι το θέμα της άμεσης αντίδρασης. Έχουμε εδώ πέρα το παράδειγμα εθνικών καταστροφών ε, που αναφέρθηκε στην Ελλάδα, στην Πολωνία και πιθανότατα θα βρεθεί και κάποια άλλη ανάλογη περίπτωση στην Ευρώπη. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι εθελοντές ε, πρέπει να προέρχονται βέβαια από διαφορετικές ε, πηγές και δεν θα πρέπει να δρουν ως πρώτη αντίδραση, γιατί η πρώτη αντίδραση συχνά ε, πρέπει να προέλθει από ανθρώπους εκπαιδευμένους και ειδικευμένους. Γνωρίζουμε το ότι η πρόληψη, η αντίδραση στις φυσικές καταστροφές βεβαίως ε, πρέπει να διασφαλιστεί και συνεργαζόμαστε και με τις εθνικές υπηρεσίες για να είναι κάπως ε, γρηγορότερες οι αντιδράσεις από τους τέσσερις μήνες και το τελευταίο είναι, ε, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το αρνούμε, είναι αυτή η υποκατάσταση της εργασίας. Και είναι η ανησυχία μας ήδη από τώρα, ε, δηλαδή να μην αντικαταστήσουν ε, εργαζόμενους οι εθελοντές. Βεβαίως το κίνητρο είναι διαφορετικό και έχουμε αυστηρές διαδικασίες και ελέγχουμε τι δραστηριότητες κάνουν ή θα αναλαμβάνουν οι εθελοντές ε, για να μην ε, είναι οι δραστηριότητες αυτές κερδοφόρες ή να μην αντικαθιστούν θέσεις εργασίας που θα έπρεπε να υπάρχουν είτε στον τομέα κοινωνικό είτε σε άλλους ε, κλάδους που καλύπτει ο τομέας της αλληλεγγύης. Αυτά από μένα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. ευχαριστώ. Ο συντάκτης γνωμοδότης, ο κύριος Ξίστοφ Χέτμαν, έχει να συμπληρώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμότατα τους συναδέλφους για τη συμμετοχή στη συζήτηση και για τις παρατηρήσεις τους. Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι όλοι συμφωνούμε ως προς την ιδέα. Και αυτό ήδη ε, είναι το ίμιση του παντός αυτή η συμφωνία επί της ιδέας και πιστεύω ότι και στη συνέχεια θα καταλήξουμε στη συμφωνία. Είμαι πολύ αισιόδοξο. Γιατί δεν άκουσα καμία αρνητική παρατήρηση που να καταδεικνύει σημαντική διάσταση απόψεων. Θα συζητήσουμε ως προς λεπτομέρειες τις επιμέρους διατάξεις. Πάντως είμαι ανοιχτός στη συζήτηση και διαλλακτικώς θα συζητήσουμε την κάθε ε, πρόταση. Αλλά η υπερβολική διευκρίνηση σημαίνει περισσότερες λέξεις, ε, περισσότερες σελίδε. Μην ξεχνάτε ότι πολλοί είναι οι δικαιούχοι που θα διαβάσουν αυτό το έγγραφο. Καλό θα ήταν λοιπόν ε, να μην πολλαπλασιάζουμε τα κείμενα, γιατί εδώ και χρόνια ζητούμε απλούστευση και περιορισμό στα ουσιώδη. Να μην ε, διευρύνουμε λοιπόν υπερβολικά την γνωμοδότηση. Πάντως ε, και για το θέμα και τη συμπληρωματικότητα προς, το, προς την εθελοντική υπηρεσία νομίζω ότι είναι σαφές ε, από την πρόταση. Εν πάση περιπτώσει θα εξετάσουμε και άλλες τροπολογίες σχετικές. Τώρα το θέμα το οικονομικό που έδειξε η κυρία Νταμάτο και είπατε, σε καμία περίπτωση να μην υποκαταστήσουν οι θελοντές ε, την απασχόληση και να μην γίνουν ένα πρόσχημα για φθηνό εργατικό δυναμικό. Ε, πολύ σωστά μας το παρουσίασε και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ε, αντιλαμβάνομαι και το θέμα το χρηματοδοτικό και το οικονομικό. Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ τα επιχειρήματα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το λόγο αυτό μεταξύ των δύο συνιστοσών του εθελοντισμού το 80% και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 20%. Εγώ πρότεινα αλλαγή του, του λόγου από 80 σε 20 σε 70-30 και σας εξήγησα γιατί. Κατά τη γνώμη μου αυτή η πρόταση έχει συμβολικό χαρακτήρα. Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμη μικρότερη διαφορά μεταξύ των δύο συνιστοσών. Αλλά συμβολικά είπα να αυξήσουμε κατά 10% το σκέλος που αφορά τη δημιουργία θέσεων, θέσεων απασχόλησης. Γιατί αυτό είναι ένα σύμβολο, είναι ένα σήμα, ένα μήνυμα προς τους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη είναι μηχανισμό για ευθυνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε ένα τέτοιο μήνυμα. Αλλά θα πρέπει να δείξουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι για μα το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό. Και σε κάθε μηχανισμό που έχουμε, σε κάθε εργαλείο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζουμε ηχηρά ότι θέλουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόληση κυρίω για τους νέους. Και αυτό είναι ένα σύμβολο, μια συμβολική χειρονομία προς τους νέους. Και θέλω να αποφύγουμε εσφαλμένες εντυπώσεις για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Σε καμία περίπτωση να μην εκλειφθεί ως μηχανισμό για τον εφοδιασμό με φθηνό εργατικό δυναμικό. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα με τον Διευθυντή, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι σίγουρα στις θεομηνίες, στις φυσικές καταστροφές, πρώτα θα πρέπει να επεμβαίνουν οι, οι ειδικευμένε υπηρεσίες της κάθε χώρας, οι εκπαιδευμένοι, οι ειδικοί. Αυτοί θα πρέπει να είναι αυτοί που πρώτοι καταφθάνουν τη στιγμή της καταστροφής ή της θεομηνίας. Αλλά μην ξεχνούμε ότι σε περιπτώσεις όπως είχαμε στην Ελλάδα με το σεισμό ε, ή με τον τυφώνα σήμερα στην Καραϊβική ή ε, την καταστροφή που είχαμε στην ε, Πολωνία ή τον καταστροφικό σεισμό στην Ιταλία. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι τα σπίτια δεν τα φτιάχνουν ούτε ειδικευμένε υπηρεσίες, ούτε οι πυροσβέστες. Τα σπίτια α, τα φτιάχνουν τοπικέ κοινωνίε. και δεν θα πρέπει αυτό να γίνεται εις βάρος της τοπικής κοινότητας και των ήδη ε, πληγή θυμάτων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κινητοποιήσουμε νέου που μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, τους πληγέντες από τις καταστροφές. Και έδωσα το παράδειγμα της Ελλάδας με το σεισμό και της Πολωνίας. Γιατί έκρινα ότι ήταν η στιγμή που θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ίσως στην Ελλάδα είναι λιγότερο το πρόβλημα και συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν εννοώ ότι είναι ε, ε λιγότερο σημαντικό. Αλλά πραγματικά αν φτάσουν μόνο το Φεβρουάριο του χρόνου οι εθελοντές, τότε είναι πολύ αργά. Άλλωστε σε μερικές ευρωπαϊκές περιφέρειες ήδη από τον Νοέμβριο αρχίζει ο χειμώνας. Οπότε και φυσικά θα πρέπει να δεσμεύσουμε και τις περιφερειακές αρχές για να το εξασφαλίσουν. Αλλά όσο πιο γρήγορα μπορούμε να κινητοποιήσουμε το σώμα αλληλεγγύης, τόσο το καλύτερο. Γιατί τότε θα δουν οι πολίτες πόσο μεγάλη προστιθέμενη αξία είναι η βοήθεια των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που φτάνουν στην πρώτη γραμμή. Και δεν έχω καμία αφιβολία για τη σημασία αυτή. Αλλά συμφωνώ απόλυτα ότι σε περίπτωση θεομηνίας πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταφθάνουν οι εκπαιδευμένοι, ειδικά εκπαιδευμένοι και οι ειδικέ υπηρεσίες. Αλλά αργότερα όταν θέλουμε να ενισχύσουμε με τους ε, νέους ε, τις κοινότητες, ε, τότε θα πρέπει να μπορούμε το συντομότερο δυνατό να τους κινητοποιούμε για να μην χρειάζεται να περάσει τόσο μεγάλο διάστημα. Και γι' αυτό είπα ότι θέλω να συνεχίσω ως προς αυτό τις συζητήσεις και τις προτάσεις. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε. Το συγκεκριμένο εργαλείο και η συμπληρωματικότητα προς την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Πολύ σημαντικό εργαλείο είναι και το Ευρωπαϊκό Σώμα για να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι σημειώσατε το πάθος της εμπλοκής σας στην υπόθεση αυτή και όπως είπατε νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα γίνει αντικείμενο μιας ευρύτερης συνένεσης ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες. Το τελικό χρονοδιάγραμμα δεν είναι ακόμα γνωστό, δεν έχει αποφασιστεί από την Επιτροπή Πολιτισμού Το θέμα λοιπόν δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Σχετικά με τη δική μας επιστροπή, εφόσον συμφωνείτε, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 14η Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Καλώς, σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Έχετε όλοι πάρει μια περίληψη των αποφάσεων αυτών. Νομίζω ότι μπορούμε να τις εγκρίνουμε διευκρινίζοντας, και το έχω ήδη πει νομίζω, ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κυκλώνα Ήρμα θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα στην Ολομέλεια. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση να θέσετε. Λοιπόν, ήταν μεγάλη χαρά για μένα που προείδρευσα. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ την επιμελητία και τη διευμηνία και όλους όσους πήραν μέρος και έδειξαν ενδιαφέρον ε, στην ποιοτικέ μας συζητήσεις. Η επόμενη συνάντηση είναι η 9η Οκτωβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 και την 3η 10 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 στις Βρυξέλλες. Καλησπέρα σας.